Bene. Allora possiamo Μπορούμε να αρχίσουμε με την πρωινή μας συνεδρίαση. Έχουμε μία μικρή καθυστέρηση. Ήλπιζα να είμαστε περισσότεροι. Αρχίζουμε με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σε σχέση με την έγκρισή της. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη χωρίς αλλαγές. Όπως ήδη ελέγχθη, θα ήθελα να σας πω ότι η συνεδρία της 21ης Φεβρουαρίου ε, ακυρώθηκε. Γι' αυτό οι ψηφοφορίες θα γίνουν σήμερα στις 4 το απόγευμα και στις 5.30 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Έχουμε δύο εκθέσεις, την έκθεση Chichester και Κέλλη. Τα πρακτικά του της 28-29 Νοεμβρίου και 17-18 ε, Δεκεμβρίου βρίσκονται στους φακέλους σας. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει κάποια υπόδειξη, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Αρχίζουμε λοιπόν με το συμπληρωματικό πρόγραμμα έρευνας για το έργο ΙΤΕΡ και δίνω το λόγο στο συνάδελφο Ρέμεκ για να μας ε, το παρουσιάσει για πέντε λεπτά. Έχουμε συνολικά 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο ομιλίας. Γίνονται ζωηρές συζητήσεις ε, για τον προϋπολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα ήθελα πέραν τούτου να σας πω ότι η ανθρωπότητα πάντα χρειαζόταν για την επιβίωσή της την ενέργεια και όλο ένα και περισσότερο και τίποτα δεν θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον. Πρόκειται λοιπόν για ένα στοιχείο κλειδί για την ίδια την ύπαρξή μας και για το μέλλον μας, δηλαδή το να επιτύχουμε επαρκή, επαρκής πηγές ενέργειας. Το ζήτημα είναι πώς θα το καταφέρουμε. Θα πρέπει να ερευνήσουμε νέες πηγές ενέργειας και η σύνδεξη είναι μια πολύ σημαντική πηγή προς αυτή την κατεύθυνση. Προτείνω ορισμένες ε, ιδέες και κάνω παρατηρήσεις που δεν είναι μόνο δικές μου. Το πρόγραμμα σύνδεξης ε, το ε, υποστηρίζει και το πρόγραμμα ίτερ. Αυτό που έχει σημασία είναι η χρηματοδότηση στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και όπως έχουν τα πράγματα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη χρηματοδότηση για δύο λόγους. Για να μην χάσει τον έλεγχο του προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για να μπορέσουμε να έχουμε την εμπιστοσύνη των ε, διεθνών εταίρων. Αυτό αφορά την έγκριση του προγράμματος ITER. Είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Ρέμεκ. Θα ήθελα να ρωτήσω ε, τη συνάδελφο Γκαρντίνη αν ε, είναι έτοιμη να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που δεν ε, άκουσα την αρχή. Λοιπόν, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία, γιατί δεν είχα ακόμα τέτοια ευκαιρία, ε, να ευχαριστήσω λοιπόν για τη δυνατότητα που μου προσφέρθηκε να αντικαταστήσω τον συνάδελφο Αλμπερτίνη ως σκιώδη εισηγητή για αυτή τη σημαντική εργασία. Να ευχαριστήσω επίσης τον εισηγητή για την εργασία που έκανε. Θεωρώ πω το κείμενο αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείο κίνηση για το οποίο ε, θα μπορέσουμε να εργαστούμε επικοδομητικά. Ε, νομίζω πως το ίτερ είναι ένα σημαντικό παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας που έχει εδρεωθεί διαχρονικά. Είναι ένα πρόγραμμα αριστείας που ενσωματώνει την έρευνα, την τεχνολογία και την ε, μηχανική αλλά και την ε, βιομηχανία του τομέα. Είμαι πεπισμένη πως η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τον κεντρικό ρόλο που έχει κατακτήσει με την υλοποίηση του ΙΤΕΡ στην επικράτειά της και ότι πρέπει σίγουρα να εγγυηθούμε την επιτυχία αυτής, αυτού του εγχειρήματο. Το ΙΤΕΡ είναι ένα πρόγραμμα που όχι μόνο πρέπει να θέσει τις βάσεις για την οικοδόμηση ε, ε, εγκαταστάσεων ε, επίδειξης αλλά και να μορφώσει, να εκπαιδεύσει επιστήμονες για αυτήν την ε, γιγάντια προσπάθεια όπου η Ευρώπη θέλει να κρατήσει την ηγετική θέση. Το ΙΤΕΡ έχει ε, συμφωνηθεί, έχει υπάρξει συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές και αυτό σημαίνει πως τα κρατημέλη θέλουν να επενδύσουν στο πρόγραμμα αυτό η συμφωνία που προβλέπει την δέσμευση 2.750 εκατομμυρίων ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον τομέα της ενέργειας. Δεν νομίζω πως είναι πια ακόμα η κατάλληλη στιγμή για να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά κάποιες ε, λαβές θα ήθελα να σας δώσω σε σχέση με το ποιο ήταν ο δικός μου προβληματισμός και η εργασία που έκανα εφόσον ε, ήρθα και λίγο αργότερα από τους συναδέλφους. Για παράδειγμα, όσον αφορά το άρθρο 3, <clears throat> συμφωνώ για τις ε, τροπολογίες του εισηγητή και ίσως θα ήταν καλό να διευκρινίσουμε κάπως περισσότερο μερικά πράγματα, όπως για παράδειγμα να περιοριστούν πάνες στα προβλεπόμενα όρια. Θα ήθελα δηλαδή να τηρηθούν οι προβλέψεις του προϋπολογισμού, γιατί πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση όπου έχουμε στους προϋπολογισμούς τέτοια προσπάθεια ε, και έχουμε ένα σωρό περικοπές, θα είναι σημαντικό να αποφύγουμε να ξεπερνάμε τον προβλεπόμενο προπολογισμό. Εξάλλου, μέσα στις προθεσμίες αυτές, ίσω να ήταν ε, απαραίτητες άλλες διευκολυνσει και αναφέρομαι για παράδειγμα στο FAST, ένα πρόγραμμα το οποίο προετοιμάζεται για να ε, μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις επιστημονικές, ε, τα επιστημονικά πορίσματα του Twitter και επίση το FAST μιλά και ασχολείται με χρήσιμε προβλέψεις όσον αφορά τις επιδείξεις. Αυτά λοιπόν έχω να πω γιατί νομίζω πως ούτως ή άλλως μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ κυρία Γκαρντίνη, η αλλως μακρηγορησα σας ευχαριστω κυρια γκαρντινη η ο συνάδελφος Ντοκάμπος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το ίτερ αποτελεί μια ευκαιρία για την βιομηχανία, για την μηχανική και για την κατάρτιση υψηλού επίπεδου στα θέματα ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι μια ευκαιρία για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων στην ίδια γραμμή λοιπόν με τις πολιτικές μας προτεραιότητες πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το ίτερ. Δεύτερο θέμα είναι αν το ίτερ πρέπει να χρηματοδοτηθεί μέσα στο πολιετές ε, ε, πλαίσιο ή όχι. Η απάντησή μας είναι ναι. Θεωρούμε και στηρίζουμε την ένταξη του Ίντερ στην πολιτική χρηματοδότηση. Πέρα τώρα από τα μέτρα, τα δημοσιονομικά και τη δημοσιονομική πειθαρχία που επικρατεί, είναι ένα, ένα τέτοιο πρόγραμμα, τέτοιες φύσεις που περιέχει τεχνολογικό κίνδυνο, είναι πιθανόν να δούμε ε, απομάκρυνση από τους, τις δημοσιονομικές του προβλέψεις. Άρα και άλλα προγράμματα όπως το ορίζοντας 2020 μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο γιατί ε, υπάρχουν εκεί τέτοια δημοσιονομικά πλαίσια που να επιτρέπουν την νομική βεβαιότητα. Πρέπει λοιπόν το ΙΤΕΡ να χρηματοδοτηθεί από τον κοινοτικό προπολογισμό, αλλά και ο ίδιος αυτός ο προπολογισμό, μάλλον η χρηματοδότηση να είναι εγγυημένη από τον κοινοτικό προπολογισμό, πέρα δηλαδή από τον τίτλο 1α, που να δίνονται εγγυήσει όπω για άλλα προγράμματα που δεν υπάρχουν μέσα, που δεν περιλαμβάνονται στον τίτλο 1α. Αυτή η πρόταση ε, θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο στην έκθεση του ε, Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεκάμπος, ο συνάδελφος Κοζανόφσκι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ υποστηρίζω πλήρως την άποψη του εισηγητή. Είναι ένα θέμα κρίσιμο και βεβαίως ε, σημαντικά είναι και τα επιχείρηματά μας. Θα ήθελα να υποστηρίξω όσους είπαν πριν από μένα πως το ίτερ είναι ένα από εκείνα τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία πραγματικά ταιριάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν το πρόγραμμα αυτό να χρηματοδοτηθεί από ένα κράτος μέλος. Είναι πολύ απαιτητικό και επιστημονικά και οικονομικά. Γι' αυτό πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα από τα κύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θεωρώ πως είναι σημαντικό να αποτελέσει τμήμα του πολιετούς ε, πλαισίου. Ένα άλλο επιχείρημα θα μπορούσε να είναι πως θέλουμε να προγραμματίσουμε επί σειρά ετών για να υπάρχει μια εγγυημένη σταθερότητα και στην επιστημονική και στην οικονομική πλευρά, όπως αξίζει το πρόγραμμα. Εγώ λοιπόν στηρίζω πλήρω τον εισηγητή και αναμένω πραγματικά να δω το πρόγραμμα αυτό να α, ε, εδρεωθεί πλήρως μαζί με το Γαλλίο και τα υπόλοιπα. Συνάδελφος Μετζάρος. Ε, σας ευχαριστώ. Υποστηρίζω τα όσα είπε η κυρία Καρδίνη και ο κύριος Τωσανόφσκι. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία και συμφωνώ με το μεγαλύτερο κομμάτι της έκθεσης. Είναι πολύ σημαντικό σημαντικό να συνεχιστεί η έρευνα. Θέλουμε να, να ζητήσουμε ε, ε, ενεργειακές πηγές και φυσικά υπάρχουν ένα σωρό δυνατότητες και σε άλλους τομείς πέρα από την, ε, πέρα από την σύνδεξη όπως η κβαντική ενέργεια. Άρα λοιπόν τα χρήματα που επενδύονται εκεί είναι πολύ σημαντικά. Και έπειτα πρόκειται, θέλουμε μάλλον να ληφθούν υπόψη τα διάφορα σχόλια που έχουν γίνει ε, σε σχέση με το πρόγραμμα έρευνας και το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, διότι το ΙΤΕΡ προσφέρει θετικά στοιχεία. Ακόμα και αν υπάρχουν κίνδυνοι, μακροπρόθεσμα η σύνδεξη θα πρέπει να ε, χρησιμοποιηθεί και ε, γιατί αυτό θα ενισχύσει τις δυνατότητές μας και την ανταγωνιστικότητά μας. Θα μπορούσαμε να ε, χρηματοδοτήσουμε το ίτερ εκτός ε, του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή φτιάχνοντας ένα συγκεκριμένο κονδύλι, αυτό θα ενίσχυε την αξιοπιστία και την βεβαιότητα των εταίρων μας και θα πρέπει να διευκολυνθεί η διεθνή συνεργασία και όχι να δυσχερεθεί. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Καρβάλιο. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με τους συναδέλφους. Το ίτερ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το μεγαλύτερο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που προωθεί η Ευρώπη, περιλαμβάνει εταιρείε, πανεπιστήμια και είναι σημαντικό να συνεχιστεί για τις αξίες των και τις τιμές εδώ πέρα το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ε, πρόταση της Κομισιόν τα 2,7 δισεκατομμύρια. Το ερώτημα λοιπόν που έχουμε είναι πού θα πάει ο προϋπολογισμός αυτός. Στα συμπεράσματα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι σαφώς στο 1α. στις προηγούμενες εκθέσεις μας και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στην ε, έκθεση που κάναμε εδώ στην Επιτροπή μας. Βάλαμε το ίτερ εντό του προπολογισμού της Ένωσης γιατί υπάρχει συνένεση πως πρέπει να υπερασπίσουμε το, τον ενιαίο ευρωπαϊκό προπολογισμό αλλά είναι πάνω από την οροφή του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου οπότε είναι εκτός του 1α Οπότε υπάρχει το πλεονέκτημα ότι αν ξεπεράσει το κόστος ε, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τα λεφτά από το 1α. Οπότε προστατεύουμε τα άλλα έργα του 1α, τον ορίζοντα 2020, το κόσμος και το Γαλιλαίο. Ή, εάν μείνει εντό του 1α, λέμε πως υπάρχει ένα υποπλαφόν, αν θέλετε, κατά τρόπον ώστε να μην επηρεαστούν τα υπόλοιπα έργα εντός του 1α. Αυτό λοιπόν σχετίζεται και με τις διαπραγματεύσεις ε, του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου και θα παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις ε, αυτές για να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε και τον ορίζοντα 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Καρβάλιο Μπαλτσούτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την σημαντική του πρόταση και θεωρώ πως ο βασικός μας στόχος σήμερα είναι να συνεχίσει να υφίσταται αυτό το έργο. Προσπαθούμε εδώ και χρόνια να βγούμε από την οικονομική κρίση. Και το ότι δεν υπάρχει κοινή ενεργειακή πολιτική εξακολουθεί να είναι πρόβλημα. Και εκτιμούμε πως ο αντιδραστήρας αυτός ε, του Ίκτερ είναι ένα νεοποιωτικό βήμα γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχίσει το έργο αυτό επιπλέον πρέπει να συμφωνήσουμε πως το πλαίσιο των ερευνητικών ε, εργασιών να μπορεί να ανακαλυφθούν ξανά να ανακαλυφθεί ξανά κάποια παλαιά σοφία και μόνο με τέτοια μέτρα θεωρώ πως θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ε, συνέχεια που είναι αναγκαία στην οικονομία. Συμφωνώ λοιπόν και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ, Ριγέρα Μαδουρέλ. Sí, muchas gracias. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, εισηγητή και θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μας ε, προσδίδει μεγάλη σημασία στο πρόγραμμα ITER και το, αυτό το ανέφεραν και προλαλήσαντες μεταξύ των οποίων ε, κυρία Κορέια. Όπως είπε η η Καρβάλιο και η Κορέιρα, το θέμα αυτό σχετίζεται άμεσα με τον προϋπολογισμό και τις ε, επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Σύμφωνα με αυτά που προείπαμε στην Επιτροπή, θα ήταν σκόπιμο τονίσουμε, όπως το έκανε και η κυρία Καρβάλιο, ότι αυτό που έχει σημασία είναι η θέση του προγράμματος στις επόμενες ε, ε, δημοσιονομικές προοπτικές που θα πρέπει να είναι εκτός του κεφαλαίου 1α για να μην έχουμε ολίσθηση ε, προς το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και γιατί έτσι θα είχαμε στη διάθεσή μας μία επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την έρευνα. Έτσι θα κέρδιζε και το σχέδιο, θα προστατεύαμε τον ορίζοντα 2020 και αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στο, στην έκθεση και εμείς θα υποβάλουμε μία τροπολογία. Ευχαριστούμε. Έλερ. Θεωρώ πως πρέπει όχι μόνο να επαναλαμβάνουμε πως το ίτερ είναι πραγματικά αποφασιστική σημασία γιατί αποτελεί μία από τις ελάχιστες τεχνολογικές εναλλακτικέ λύσεις, αλλά είναι και ένα ερευνητικό πρόγραμμα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την, ε, τις τεχνικές δυσκολίες, γιατί υπάρχουν αυτές και είναι ένα πολύ μακρόπνο σχέδιο και μπορεί επειδή είναι ερευνητικό έργο να γίνει ακόμη πιο ακριβότερο. Αλλά βεβαίως αυτό προϋποθέτει και πρέπει να το πούμε αυτό, ε, σοβαρή ενασχόληση με το ίτερ. Τα τελευταία χρόνια είχαμε καταστροφική διαχείριση, είχαμε ερωτήσεις από τη βιομηχανία για το τι γίνεται με τις δημόσιες προμήθειες, είχαμε μια δομή που είναι συμβιβαστική αλλά δεν έχει ουδεμία σχέση με αποτελεσματική διοίκηση. Δηλαδή βρίσκεται το ίτερ στην Νότια Γαλλία, η διοίκηση στην Ισπανία η συνεργασία μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών που τίθεται ένα αμφιβόλο αν δει κανεί τα αποτελέσματα. Οπότε ε, υπάρχουν κάποια διέξοδα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε. Και πρέπει επίσης να πούμε τώρα πως κάθε χρηματοδότηση του προπολογισμού που είναι κάτω από 4 δισεκατομμύρια είναι αστεία. Έχουμε αυτή την δέσμευση από τις διεθνείς συνθήκες ανεξαρτήτως του, τι, ε, του πώς εξελίσσεται η οικονομική κατάσταση. Αν λοιπόν δεν γράψουμε κάπου στον προπολογισμό αυτά τα 4 δισεκατομμύρια, πρέπει να το ξέρουμε πως θα έχουμε μετά υπερβάσεις. Είναι ανεπαρκής η πρόταση του Συμβουλίου, 2,7 δισεκατομμύρια δεν είναι εγγύηση, τα 4 είναι εγγύηση του κόστους. Και είχαμε τον ε, συμβιβασμό του προγράμματος ε, πλαισίου 7, πως επειδή είναι ερευνητικό ε, έργο, αν έχουμε υπερβάσεις θα πάνε σε άλλο τίτλο. Και το μίνιμουμ είναι 4 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε. Αν κάνουμε κάτι τέτοιο πρέπει να ξέρουμε πως θα κανιβαλίσουμε άλλα έργα στην επόμενη προγραμματική περίοδο για να βρούμε τα λεφτά. πρέπει να μπουν κάπου στον προπολογισμό τα 4 εκατομμύρια. Δεν έχει νόημα να ελπίζουμε πως κάπου μέσα στο 1α θα βρεθούν λεφτά. Χρειαζόμαστε ένα προπολογισμό 4 δισεκατομμυρίων που θα είναι σίγουρος και δεν γίνεται αυτό μέσω του 1α. Grazie al collega la parola al Andrea. Ο κύριος Καρινιάνη έχει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής. Άκουσα με προσοχή όλα τα σχόλια και θα ήθελα να πω κάτι το σημαντικό για την Κομισιόν και αυτό το ε, ανέφερε ο Επίτροπος στο ε, Συμβούλιο ε, πρόσφατα. Η συγκράτηση του κόστους έχει μεγάλη σημασία. Αυτό αναφέρθηκε και στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Και αυτό αφορά και την παρουσία της Euratom στην διακυβέρνηση, στη διαχείριση του ΙΤΕΡ. Αυτό το αναφέραμε πρόσφατα και στους ε, διεθνείς εταίρους μας. Άρα, όπως ήδη ελέγχθη, έχουμε αναλάβει μία διεθνή δέσμευση αλλά έχουμε 6,6 δις και πολύ μεγάλες ε, δηλαδή περικοπές και δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, προσθήκες εκτός και αν αυτό είναι αναγκαίο γιατί δεν μπορούμε να καταβάλουμε επιπρόσθετο κόστος. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Ρέμεκ, ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που παρουσίασαν τις απόψεις τους. Εγώ θα δεχτώ αυτές τις υποδείξεις. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τους ε, πάντες και νομίζω ότι η η συνεργασία αυτή θα οδηγεί στην υπέρβαση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ριβάζη θέλει το λόγο για ένα λεπτό. Είναι σκιώδης από τους πράσινους. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι μας φοβίζει το γεγονός ότι το κόστος της ε, γης έχει, των γεών έχει αυξηθεί επί τρία. Στο μεταξύ θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη σε εκούσια βάση, σε θελούσια βάση θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν το ίτερ γιατί οι Άγγλοι με το JET ή οι Γερμανοί έχουν το δικό τους ε, πρόγραμμα σύνδεξης βεβαίως δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε και τα 6,6 δις που είναι η συνεισφορά των κρατών μελών. Ως επιστήμων βρίσκω ότι στην πρόταση ψηφίσματος δεν προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλους τους, τους επιστήμονες για το ίτερ για να δούμε πού υπάρχουν χάσματα για την ε, κατασκευή του διότι στον προϋπολογισμό μιλάμε μόνο για χρήματα και όχι για μελέτη ε, σκοπιμότητας. Όταν μιλάμε για την ηλεκτρική ενέργεια το 2005 και επειδή το ίτερ ε, ε, θα ασχοληθεί μόνο με την δημιουργία και παρασκευή πλάσματος και όχι ενέργειας, θα χρειαζόμαστε να βρούμε νέες πηγές το αργότερο μέχρι το 2100. Δεν ξέρω λοιπόν ε, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Όταν βλέπουμε ε, χώρες όπως την Ελλάδα και άλλες χώρες, δεν βλέπω πώς μπορούν να συμμετάσχουν. Εξαιρετική η ενέργεια, ε, μιλάμε για ανανεώσιμες, είναι εφικτό, αλλά εδώ δαπανούμε χρήματα χωρίς να έχουμε καμία επιστημονική εγγύηση. Και τέλος, στο Κανταράς ζήτησα ως ε, ευρωβουλευτής να συμμετάσχω, αλλά μου το αρνήθηκαν γιατί το ίτερ δεν επιτρέπει καμία επικριτική νότα. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα γίνει στη συνέχεια αν δεν έχουμε ε, πρόσβαση στις πληροφορίες σε σχέση με τη βέλτιστη δυνατή χρήση. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους, λέει η Πρόεδρος, ότι έκανα ε, εξαίρεση αυτή τη φορά για την κυρία Ριβάζη, αλλά δεν θα ξανανοίξω τη συζήτηση. Τώρα βεβαίως ο κύριος Ρέμε ξαναζήτησε το λόγο για να απαντήσει στην κυρία ε, Ριβάζη του δίνω το λόγο, αλλά δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όταν έχει κλείσει η συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σε σχέση με την τελευταία παρέμβαση θα ήθελα και εγώ να λάβω το λόγο διότι πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει συγκεκριμενοποίηση σε πολλούς τομείς, αλλά όχι σε αυτόν. Ε, σας ομολογώ ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία έρευνας και εξερεύνησας, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία λειτουργεί, υπάρχει, προϋπάρχει στη φύση. Η σύνδεξη ε, αποτελεί κινητήρια δύναμη της φύσης λειτουργεί για τον ήλιο, υπάρχει για τον ήλιο και γι' αυτό έχουμε εκατό, εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια όπου βλέπουμε ότι, διαπιστώνουμε ότι λειτουργεί η σύνδεξη και βλέπουμε πώς λειτουργεί η σύνδεξη και σε χώρες όπως η Γερμανία. Στο Κάλαμ είδαμε πώς λειτουργεί το ολοπλαίσιο και πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές οι έρευνες είναι πολύ σημαντικές. Νομίζω λοιπόν ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ξανανοίξουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ τον κύριο Ρέμεκ και τώρα Ανοίγει η φάση των τροπολογιών. Οι τροπολογίες λοιπόν πρέπει να κατατεθούν εντός της 28 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Επόμενο σημείο της της διάταξης για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Ο συνάδελφος Μπούζεκ έχει το λόγο. Ε, Μπούζεκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή μου σήμερα να είμαι ο εισηγητής για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Είναι κάτι το σημαντικό και επειδή είναι τμήμα της ε, Δεύτερη νομοθεσία περί ενιαία αγοράς είναι και ένα τομέα προτεραιότητα. Αν θέλουμε να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά πρέπει να ξεκινήσουμε από την ενιαία αγορά ενέργειας. Είναι μια προτεραιότητά μας για να ξαναυπάρξει οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δημιουργώντας την αγορά αυτή μπορούμε να περάσουμε στην στρατηγική του 2020 και τις συνθήκες για να ξεπεράσουμε την κρίση. Και αυτό είναι σημαντικό. Να πω τη γενική μου άποψη σε τέσσερα σημεία. Αλλά και να τοποθετηθώ για ως προς την ανακοίνωση της Κομισιόν. Πρώτον λοιπόν, πώς θα πρέπει να δημιουργηθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας, όπως ε, ισχύει και για την ενιαία αγορά για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, έτσι και η αγορά της ενέργειας πρέπει να προσανατολίζεται στους πελάτες, είναι προφανές. Πρέπει να δημιουργηθεί με τρόπο ε, παρόμοιο όπως η αγορά για τα αγαθά και τις υπηρεσίες πριν από κάποιες δεκαετίες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να είναι ανοιχτή για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Με ε, αξιόπιστη ε, πάροχη ενέργειας με καλύτερο συντονισμό των αγορών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο, σημαντικό, πρέπει να είναι ανταγωνιστική και να δημιουργεί ανταγωνισμό και πιθανώς και χαμηλότερες τιμές ενέργειας να υποστηρίζει τη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και βεβαίω έχουμε και τον ορίζοντα 2020, το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο, όλα αυτά τα ενεργειακά έργα. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει και σωστή ρύθμιση. Δεν είναι εύκολο, αλλά κάτι τέτοιο προτείνουμε. Το προτείναμε πριν από τέσσερα χρόνια. Ήταν το τέταρτο ενεργειακό πακέτο που ολοκληρώθηκε το 2009 με προθεσμία εφαρμογή στο Μάρτιο του 2011 και μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί από πολλά κράτη-μέλη. Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και για να σταματήσει η κρατική παρέμβαση στις τιμές ενέργειας. Όπως δεν συμβαίνει σε 18 κράτη-μέλη. Οπωσδήποτε είναι το πιο ε, πρόβλημα, αλλά βεβαίω ε, η απόφαση επαφείεται στα κράτη-μέλη και η ευθύνη μας σήμερα είναι να τους υπενθυμίσουμε πως η υποχρέωσή τους είναι σαφής. να εφαρμόσουν δηλαδή όλα όσα λέει το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Και τέλος, πώς πρέπει να δημιουργήσουμε μια τέτοια αγορά. Πρέπει να υπάρχει διασύνδεση ε, των δικτύων ε, με την ε, απαραίτητη συμβατότητα, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει η πλήρης διασύνδεση δηλαδή των συστημάτων ε, μεταφοράς απαιτεί πολλά κονδύλια. Θα πω λίγα λόγια μετά για αυτό το θέμα. Και βέβαια υπάρχουν και ε, απομονωμένες ενεργειακά περιοχές. Κατόπιν, οι αδυναμίες μας. Η γενική κατάσταση δεν είναι ακόμα ικανοποιητική. Έχουμε ακόμα πολλά που πρέπει να επιτύχουμε. Ε, ξεκινήσαμε πριν από μια δεκαετία με τον λεπτισμό, ε, το φυσικό αέριο και διάφορες οδηγίες και προτάσεις. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο σοβαρές ε, αδυναμίες. Πρέπει να τα πούμε αυτά στην έκθεση και να στηρίξουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει μια απόφαση για να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες. Περισσότερες επενδύσει στον τομέα αυτών βασίζονται σε επιδοτήσεις. Γιατί βεβαίω έχουμε εθνικές και περιφερειακές αγορές και αγορές διαφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι επαρκώς ανοιχτέ. και έτσι δεν μπορούν να μπουν με φορείς. Να δώσω κάποια παραδείγματα. Σε κάποιε περιπτώσει οι τιμέ φυσικού αερίου είναι τέσσερι φορές υψηλότερες από αλλού. Γιατί όπως είπα είναι απομονωμένες οι αγορές. Σε κάποια μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο ασφάλειας είναι πολύ χαμηλότερο από αλλού. Σε πολλά κράτη-μέλη οι καταναλωτές ε, δεν έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν ε, εταιρεία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα. Δεν είμαστε αποτελεσματικοί στο να κάνουμε επενδύσει στην ε, αποτελεσματική χρήση ενέργειας, συμπαραγωγή ενέργεια, ε, παραγωγή από ΑΠΕ. Γιατί, γιατί δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες για την αγορά. Δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα, κανόνες εμπορικοί. Τώρα ξεκινήσαμε μόλις με τα σχετικά πιστοποιητικά. Αλλά δεν έχει τελειώσει βεβαίως αυτή η υπόθεση που έχουν πολλά να γίνουν ακόμα. Πρέπει λοιπόν να επισημάνουμε στην έκθεσή μας όλα αυτά τα πράγματα και βεβαίως ε, πρέπει να τονίσουμε και τα πλέον εκτήματα όχι μόνο τις ε, αδυναμίες πιθανώ καλύτερε τιμέ, καλύτερο έλεγχο του κόστου της ε, ενέργειας, 13 δισεκατομμύρια ευρώ για τους ευρωπαίου καταναλωτέ θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν ετησίω. χάρη στην ενιαία αγορά. Και βεβαίως ε, ε, θα, προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσουμε νέες θέσει εργασίας γιατί υπάρχει μια αγορά για 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Μια φανταστική αγορά και βεβαίως θα έχουμε και υψηλή τεχνολογία και σημαντικότερο και για τις γενικότερες σχέσεις Ένωσης. Θα έχουμε δηλαδή ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση απέναντι σε εξωτερικούς προμηθευτές εάν ε, συντονιστούμε στις αγορές μας. Και βεβαίως δεν θα έχουμε διακοπές και λήψεις και τα λοιπά. Και τελευταίο, τι πρέπει να γίνει μέχρι το 2014. Να τελειώσω. Μία πρόταση που είχε γίνει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, το 2011. Και ε, ε, το 2010 ήταν οι επενδύσεις 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου ενέργειας, ελαχιστοποίηση των ε, διαφορών μεταξύ κρατών μελών και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο. Κάποια από αυτά τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται ε, επαρκώς από την ανακοίνωση της Κομισιόν και θα ήθελα να πω αυτό πραγματικά τελευταίο ευχαρίστω να δεχτώ τις προτάσεις σας, αμφιβολίες σας κτλ. Πώς πρέπει να συνεργαστούμε και χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις και αναμένω τη συνεργασία με τους κοιόδης συγητές για να καταλήξουμε σε ένα επικοδομητικό έγγραφο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μπούζεκ. Τώρα οι συνάδελφοι σίγουρα θα με βοηθήσουν να ε, προλάβουμε το χρόνο που δώσαμε, τον παραπανήσιο χρόνο που δώσαμε στον ε, εισηγητή. Πρώτα ο συνάδελφος Ντεο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εργαζόμενος ε, εξ ονόματος της συναδέλφου Ζούντιτ Μέρκη. θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή, όχι μόνο για το όσο έχει ήδη κάνει εδώ, και δεν μιλώ βέβαια για το παρελθόν, αλλά και για το όσα είπε σήμερα. Με τα οποία συμφωνούμε σχεδόν απόλυτα. Η εσωτερική αγορά ενέργειας είναι κρογωνίος λίθος της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δημιουργεί ανταγωνισμό, ανοίγει ελεύθερη αγορά, κινητοποιεί τις πόρους ανανεώσιμης ενέργειας και ε, το μέλλον θα είναι καλύτερο όταν ο ίδιος ο καταναλωτής θα μπορεί να συνδέσει το ηλιακό του θερμοσύφωνα ο ίδιος στο δίκτυο. Ωστόσο, <clears throat> θα πρέπει να δούμε πώς θα φτάσουμε σε όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Καταρχήν, η θετική προσοχή της Κομισιόν δίνει μεγάλη σημασία στην ισχύ του καταναλωτή. Αναγνωρίζει ότι για να εκμεταλλευτούμε τα πλονεκτήματα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, οι καταναλωτές και οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν και να κινητοποιηθούν για να παίξουν ενεργό ρόλο στην αγορά. Είναι οι βασικοί παίκτες στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Στις κάτω χώρες βλέπουμε πολλές αυθόρμητες πρωτοβουλίες στις τοπικές κοινότητες και στα νοικοκυριά για να παράγουν την ενέργειά τους. Η Κομισιόν πρέπει να στηρίξει περισσότερο αυτή την τάση, κινητοποιώντας τους πολίτες ώστε να συμμετέχουν στην ενεργειακή αγορά και να μειώσει τους τα πιθανά εμπόδια σε κάτι τέτοιο. Επίσης πρέπει να στοχεύσουμε τη βοήθεια στους ευάλωτους καταναλωτές γιατί υπάρχει μια εκτίμηση ότι πάνω από 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους και να διατηρήσουν ε, άνετο βιωτικό επίπεδο. Ωστόσο, οι τιμές ενέργειας αυξάνονται διαρκώς και αυτή η μελέτη δείχνει πως οι τιμές της ενέργειας στην Ολλανδία ανέβηκαν πάνω από 50% κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι όλα ένα και περισσότερα νοικοκυριά δεν μπορούν πια να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Δεν βλέπω επαρκείς προτάσεις για μέτρα που θα πρέπει να λάβει η Κομισιόν για να στηρίξει πραγματικά αυτού του καταναλωτέ δεν είναι σαφές ε, για το ποιες, ενέργειε ενέργειες θα αναλάβει ώστε να δαρθούν νέες ανανεώσιμες πηγές. Πρέπει να Αντιμετωπιστούν επίση τι τρευλώσει τη αγορά, όπω η έλλειψη τη διαφάνεια, τα επιδοτήσει για μη φιλικές προ το περιβάλλον πηγέ ενέργεια ή μονοπόλια. Επίση πρέπει να δούμε θέματα όπω η ασφάλεια τη θεματα οπως η περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων και η επιτάχυνση των ευφυών δικτύων. Τέλος, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ολοκληρωμένη εθνική αγορά και στην ολοκληρωμένη πραγματική ευρωπαϊκή αγορά. Και είναι κρίμα που ο προπολογισμό αυτός, ο προϋπόμενος, ε, προβλέπει σοβαρές περικοπές στον τομέα της ενέργειας. Με, λόγα, με τόσο λίγα χρήματα πώς να δημιουργήσουμε μια πραγματική αγορά. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Σιμάνσκι, παρακαλώ. E, Ευχαριστώ. Ω συζητητή ε, για το Κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών θα ήθελα να πω πω σε πολλού ε, τομεί ε, τη ενιαία αγορά έχουμε δει πω είναι δυνατόν να κερδίσουμε πάρα πολλά για τους Ευρωπαίους πολίτες, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, την ευρωπαϊκή βιομηχανία και αυτό όχι μόνο από την κλίμακα των όσων συμβαίνουν, αλλά λόγω και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Εάν δούμε το τι γίνεται στον τομέα της ενέργειας, έχουμε ήδη επιτύχει πολλά. Έχουμε το τρίτο ενεργειακό πακέτο, έναν κανονισμό για την ασφάλεια της ε, προσφοράς ε, και βεβαίως έχουμε και την ε, αγορά χοντρικής η οποία θα επηρεαστεί και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις της. Αλλά ξέρουμε πως δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά της ενέργειας και για να ολοκληρωθεί επιτέλους δεν είναι αυτό κάτι το οποίο θα λυθεί μόνο με νόμους και κανόνες, πρέπει να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό. Χρειάζεται περισσότερη καταπολέμηση των μονοπωλίων γιατί εξακολουθεί να είναι βαριά ακόμα η σκιά των μονοπωλίων. Οπότε δεν είναι θέμα μόνο ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και τα όσα έχουμε ήδη επιτύχει. Πρέπει λοιπόν να δούμε το ενεργειακό πακέτο και να το προστατεύσουμε απέναντι σε ε, εκείνους τις ε, εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δηλαδή τη Ρωσία και την Κασπρόμ, που έχουν δικές τους απαιτήσει. Και προφανώς θεωρώ πως πρέπει να κάνουμε και τις απαραίτητες αλλαγές. Δεν θέλουμε να αυξηθεί η τιμή, γιατί κάτι τέτοιο θα είναι ανταπαραγωγικό αν υπερβάλλουμε με τα περιβαλλοντικά μέτρα. Οπότε πρέπει ε, να έχουμε μια ισορροπημένη εσωτερική αγορά. Μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται συχνά. Και ε, όπως είπα πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία όσον αφορά την κλιματική πολιτική. Προφανώς θα είναι επίσης επωφελές να έχουμε μια εσωτερική αγορά ενέργειας για να έχουμε κάποια αύξηση στην ε, ασφάλεια παροχής και τέλος είμαι ευγνώμων προς την Κομισιόν, γιατί αν δείτε την ανακοίνωση, βλέπουμε πως έχουν μία ανακοίνωση για την πορεία προς το 2050, αλλά προφανώς οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς πρέπει να γίνουν σήμερα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να Αμ δώσω κάποια στοιχεία για τις τροπολογίες που θα υποβάλω σε σχέση με αυτήν ε, την ε, έκθεση και που αφορούν ε, το δική μας οπτική για το πώς θα πρέπει να έχει ο τομέας της ενέργειας που είναι ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομίας για την ανεξαρτησία κάθε, κάθε χώρας αλλά και για την ανάπτυξη. Καταρχήν θεωρώ πως όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν εγγύηση και βεβαιότητα πως έχουν ενέργεια στη διάθεσή τους, ότι δηλαδή έχουν ενεργειακή και κυριαρχία και τις δυνατότητες να αναπτυχθούν μέσω αυτής της ενεργειακής κυριαρχίας. Για τον ε, πληθυσμό θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια ανεφοδιασμού, δηλαδή δεν ε, μπορούν ε, να εξαρτώνται όλα από συγκεκριμένα συμφέροντα. Θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια ανεφοδιασμού. Απ' την άλλη πλευρά θεωρώ πως ο στρατηγικός τομέας ε, της ενέργειας ε, θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία της ε, παραγωγικής διαδικασίας, παραγωγής και ανάπτυξης που τόσο αναφέρεται, δηλαδή στην υπηρεσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τον επιχειρηματικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα θα πρέπει να εξυπηρετεί η ενέργεια με υπηρεσίες και σε τιμές που να μπορούν να τις πληρώσουν. Ενώ βλέπουμε τι συμβαίνει σε πολλές χώρες γιατί η τιμές αυξάνονται σε βαθμό που δυσκολεύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά να είναι στην υπηρεσία των λαών ώστε να υπάρχει ενέργεια για όλους σε προσιτές τιμές. Όμως η ιστορία μας δείχνει πως η απελευθέρωση τομέα δεν οδήγησε σε μείωση του κόστους μέσω, μια, μέσω του ανταγωνισμού ε, σε αυτό το τομέα δεν λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο που αναμέναμε η ε, απελευθέρωση είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της χώρας μου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα ενώ μειώνονται οι μισθοί των εργαζόμενων, τα κέρδη των επιχειρήσεων ε, ενέργειας και φυσικού αερίου αυξάνονται διαρκώς. Η μονοπωλιακή εταιρεία ηλεκτρισμού κέρδισε παραπάνω 57% από ό,τι το 2011. Για φέτος η επιχείρηση καυσίμων αύξησε 6 φορές τις τιμές των καυσίμων. Δεν υπάρχει καμία λογική σε όλα αυτά. και οποιοδήποτε στόχος κοινωνικής συνοχής ή κοινωνικής δεοκίνης λείπει, απουσιάζει από αυτή την κατάσταση. Θέλουμε λοιπόν να συστήσουμε την αύξηση, την ενδυνάμωση του, του ρόλου του κράτους σε αυτή την υπόθεση και τη δυνατότητα ε, η απόδοση, η, τα κέρδη που έχει ο τομέας να ανακατανέμονται με δίκαιο τρόπο και να επιδιώκουν κοινωνικούς στόχους και όχι κέρδη για τους λίγους. Θεωρούμε πως αυτή θα ήταν μια σημαντική συμβολή στην ε, υπέρβαση της κρίσης. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει συνάδελφος Κράουσμαν που αντικαθιστά την Ρόντμπεκ. Εμείς ε, ως ε, φιλελεύθεροι τασόμαστε υπέρ της εσωτερικής αγοράς καθώς και τις σχετικές φιλοδοξίες για δημιουργία ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο θα είναι ευεργετικό για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Ε, χαμηλώνοντας τις ε, τιμές, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει και θέσεις ε, απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια της παραγωγής με χαμηλή ε, χρήση άνθρακα. Οι φιλελεύθεροι συμφωνούν με την Κομισιόν ότι ε, υπάρχουν προσκόμματα για την ε, δημιουργία ενέργεια στη στιγμή που ρυθμίζουμε την πολιτική τιμών στην εσωτερική αγορά. Αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο πρόσκομα, γι' αυτό προτρέπουμε την Κομισιόν να ρυθμίσει τις ε, ε, τιμές ενέργειας και ηλεκτρισμού για τους ε, καταναλωτές και να ορίσουμε τις ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών για να μπορέσουμε να τους ευεργετήσουμε. Ακόμα και οι ρυθμισμένες τιμές μπορούν να μην αποστέλουν το σωστό μήνυμα στην αγορά. Οι επενδυτές θεωρούν την, τον προκαθορισμό τιμών ως πολιτικό παρεμβατισμό. Η Επιτροπή υποδεικνύει στα κράτη-μέλη να ε, δημιουργήσουν εφείς ε, μετρητές και μηχανισμούς. Επίσης, η ε, ευφυείς μετρητές είναι αναπόσπαστο μέρος του προκαθορισμού αυτού τιμών, καθώς και δίκτυα και δικτύων έτσι ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η Επιτροπή επίσης τονίζει την ανάγκη για τα κράτη-μέλη να προβούν σε εξυγχρονισμό των ε, ε, δικτύων ηλεκτρισμού μέσα στα πλαίσια για το ICT. Γιατί οι διανομής έχουν κίνητρα, θα πρέπει να αποστέλουν μηνύματα κινήτρων για νέες επενδύσεις, έτσι ώστε να υπάρχει ε, ευελιξία στη χρήση των δικτύων. Είναι κρίμα που το Συμβούλιο έχει μειώσει ε, ε, τη χρηματοδότηση του μέσου Connecting Europe. Οι περικοπές αυτές, με τις περικοπές αυτές το Συμβούλιο καθιστά πολύ πιο δύσκολη την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και οι φιλελεύθεροι εκφράζουν τη λύπη τους για αυτή την απόφαση του Συμβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ, Πιλάρ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σήμερα βρισκόμαστε στην ε, απαρχή μιας συζήτησης για μια πρόταση που μας αποστέλει η Κομισιόν για να δώσουμε μια όθηση στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Είναι μια αγορά που χρειάζεται αυτή την όθηση ευρείας κλίμακας γιατί μιλάμε για 500 ε, εκατομμύρια καταναλωτές, ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο συνάδελφος ε, Μπούζεκ μας είπε, μας ανέφερε πολλά επιμέρους ζητήματα, πάντα τον ακούω με προσοχή και αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε κάπως συντονισμένοι. Θα ήθελα να ε, τα εξής. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί πυλώνες για να ε, βασιστούμε για αυτή την αγορά της ενέργειας. Μία επελευθερωμένη αγορά και μία ανταγωνιστική αγορά. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί άξονες και αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να ισχύσει και το τρίτο ενεργειακό πακέτο το οποίο να επαφείται στους δύο αυτούς άξονες. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο και θα πρέπει η Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Δύο είναι οι άξονες. Μία απελευθερωμένη αγορά και μία ε, ανταγωνιστική αγορά. Επίσης, μία αγορά με διαφάνεια και όλες τις πληροφορίες για τις ΜΜΕ και τον καταναλωτή, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να επιλέξει. Γιατί μόνο ένα τρίτο των καταναλωτών μπορούν να συγκρίνουν. Μιλάμε λοιπόν για μια πραγματική δυνατότητα επιλογής ε, μέσω μιας ε, διαφανούς και ανταγωνιστικής αγοράς με αλληλοσυνθέσεις, με δίκτυα μεταφοράς και διανομής για να διακόψουμε αυτούς τους ενεργειακούς ε, θύλακες που αποτελούν ορισμένα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη διασυνδεσιμότητας. Χρειαζόμαστε μία ανταγωνιστική αγορά, μία διαφανή αγορά και μία αγορά με δίκτυα τα οποία να είναι αποτελεσματικά για να διακόψουμε ε, αυτούς τους ενεργειακούς θύλακες που ισχύουν και στην ε, Ισπανία μεταξύ άλλων. Η κυρία Χιμπνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η υποστηρίζουμε και συμπληρώνουμε την ε, εσωτερική αγορά ενέργειας και ελπίζω να το πετύχουμε αυτό, να φτάσουμε σε μια πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας για να υποβοηθήσουμε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές και να λάβουμε υπόψη τις ε, εξατομικευμένες τους ανάγκες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε την αγορά αυτή για τη, τα αγαθά, για τις υπηρεσίες, για τον τριτογενή τομέα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στους στόχους μας. Χρειαζόμαστε ευφυή ε, ε, δίκτυα και διασυνδεσιμότητα, έτσι ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα των υπηρεσιών στον ε, ίδιο βαθμό σε όλους. Πολύ συχνά λέμε ότι οι συμβατικές πηγές ε, ενέργειας δεν είναι επαρκείς και θα πρέπει να σταθούμε στις ανανεώσιμες, να στραφούμε στις ανανεώσιμες. Χρειάζεται όμως και η χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας, αλλά θα πρέπει να διερευνήσουμε πολύ περισσότερο τις δυνατότητες που μας διανοίγονται από τις ε, ανανεώσιμες. Μέσω της έρευνας λοιπόν θα δημιουργήσουμε νέες τεχνολογίες και θα σταθούμε στις μη συμβατικές ε, πηγές ενέργειας, διότι δαπανούμε πολλά χρήματα για την ανάπτυξη νέων ε, ενεργειακών μέσων και πηγών. Οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να, ε, να αναγνωρίζουν και να γνωρίζουν καλύτερα, να μπορούν να ερμηνεύουν τους λογαριασμούς που, που παίρνουν. Γιατί δυστυχώς έχουμε μία πηγή ενέργειας και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε γιατί υπάρχει ένας προμηθευτής στην αγορά. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα εφίους μέτρησης και μία πολύ καλή ε, χρήση ενέργειας για να πέσουν και οι τιμές ενέργειας χωρίς αυτό να είναι επιζήμιο ως προς την ε, ποιότητα. Θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις δαπάνες αλλά να υπάρχει ε, διαφάνεια ως προς τις προμήθειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι πολλές φορές ε, ε, εξωγενείς φορείς επιβάλλουν και τους όρους τους στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλές δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να κατασπαταλούμε τις δυνατότητες που έχουμε. Η κυρία Κουκόβιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Γερζι Μπούζεκ για την έκθεσή του χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι ρυθμίσαμε ε, πρώτα απ' όλα τα, την κινητή τηλεφωνία. Βεβαίω και ο ηλεκτρισμός είναι κάτι το βασικό. Αλλά βεβαίω θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία μιας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι πώς, πώς θα προσελκύσουμε νέους επενδυτές, γιατί ε, αυτό θα έχει αποτέλεσμα ανάπτυξη και δουλειές. Αυτό είναι βασικό. Δεύτερον, πώς θα προωθήσουμε την έρευνα, ειδικά στο πώς θα αποφεύγουμε τις απώλειες κατά τη μεταφορά και πώς θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και από τους παραγωγούς, τους ηλεκτρικούς σταθμούς, γιατί διαφέρουν πάρα πολύ από τους παλαιούς ε, ηλεκτρικούς σταθμούς που είχαν απόδοση 30% μόνο. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε και αυτή την αποτελεσματικότητα και κατά κανόνα βέβαια χρειάζεται και κοινή έρευνα εδώ πέρα. Και πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα συμπεριλάβουμε τις ε, ανανεώσιμες ενέργειες στα συστήματα μεταφοράς ενέργειας. Γιατί υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπαλτσούτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Μπούζεκ, τον εισηγητή. Έχει ε, αναφερθεί πάρα πολλές φορές η τοποθέτησή του, η έκθεση νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους μέχρι το 2014 υποτίθεται πως δεν θα υπάρχουν ε, απομονωμένες αγορές, αλλά από δεν θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Εγώ προέρχομαι από μια γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή και Ελπίζω να έχουμε πιο γρήγορη πρόοδο από το μέχρι στιγμής. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Σχετίζονται με την ρυθμίση των τιμών της ενέργειας, το τρίτο ενεργειακό πακέτο, τα μονοπόλια κάποιων εταιριών Επίσης, μιλάμε για τη ρύθμιση των τιμών, αλλά το πρόβλημα αυτό θα λυθεί όταν θα έχουμε τις απαραίτητες ε, υποδομές. Γι' αυτό θα πρέπει να προγραμματίσουμε για την, την αποτελεσματικότητα. Π.χ. στην περιοχή της Βαλτικής είχαμε συχνά ε, ζητήσει ε, ένα, έναν ε, τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου και για τις τρεις χώρες. Και μάλιστα να γίνει κάτι τέτοιο μέχρι το 2030. Αυτό αργεί πάρα πολύ, γι' αυτό η Λιθουανία αποφάσισε να χτίσει, να φτιάξει μόνη της ένα τέτοιο, ένα τέτοιο τερματικό σταθμό. Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα λοιπόν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ Τζόρνταν. Ευχαριστώ. Τέσσερα βασικά πράγματα και απλά έχω να πω. Πρώτα απ' όλα η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν μπορεί να δουλέψει με ε, επιδοτήσεις και ρυθμισμένες τιμές. Δεύτερον, η ευρωπαϊκή αγορά δεν μπορεί να είναι ε, το άθροισμα 28 εθνικών πολιτικών. Ακόμα και η Γερμανία δεν θα υιοθετήσει μόνο τις αποφάσεις που επηρεάζουν τα μισά τουλάχιστον κράτη-μέλη. Και το τρίτο μου μήνυμα είναι πως δεν, μπορούμε να δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά με υπερβολική ρύθμιση. Αυτό προκαλεί αστάθεια. Τα μηνύματα αυτά είναι απλά, αλλά πρέπει να ε, προσαρμόσουμε 27 εθνικές πολιτικές και ευρωπαϊκή εθνική πολιτική και την ευρωπαϊκή μεσχόλητη ενεργειακή πολιτική σε αυτά τα απλά πράγματα. Αλλιώς δεν θα επιτύχουμε την κοινή ενεργειακή μας πολιτική και τέταρτο και τελευταίο η απόφαση για το πολιετές μισονομικό πλαίσιο για το να περικοπούν στο μισό τα κονδύλια του μέσου συνδέοντας στην Ευρώπη είναι απαράδεκτη. Και είναι απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που υποτίθεται αποφάσισε πλήρη εφαρμογή της ενιαίας αγοράς ενέργειας μέχρι το 2014. Ευχαριστώ, Μπένστεν. Eh, Øh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούζεκ για αυτή την ε, εξαιρετική έκθεση. Θα πρέπει να ε, μιλήσουμε για μια νέα πραγματικότητα στην εσωτερική αγορά. Αν πρόκειται να έχουμε εσωτερική αγορά δεν μπορεί να υλοποιηθεί παρά μόνο όταν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός, κάτι το οποίο δεν ισχύει τώρα. Ε, έχουμε, ζούμε καταστάσεις ε, μονοπωλίου. Έχουμε γιγάντιες επιχειρήσεις αλλά δεν υπάρχει επαρκής ε, διαφάνεια. Το... Τα δύο τρίτα των ε, χωρών ε, δεν έχουν εφαρμόσει το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης αγοράς. Γι' αυτό θα πρέπει η Επιτροπή να επιβάλλει κυρώσεις στις χώρες που δεν εφάρμοσαν το πακέτο. Στην ευρωπαϊκή οικογένεια λοιπόν χρειάζονται αυτοί οι ενεργειακοί θύλακες. Άκουσα την ε, ε, Πιλάρ να μιλάει για αυτούς τους ενεργειακούς ε, θύλακες στην Ισπανία, αλλά τι γίνεται με την Εστονία και τη Λιθουανία που καταβάλουν το διπλό αντίτιμο για το φυσικό αέριο σε σχέση με τη Γερμανία. δεν μπορούμε να δεχτούμε οι βαλτικές χώρες να καταβάλουν τέτοιο υψηλό αντίτιμο για την ενέργεια. Αυτό ισχύει και για το ε, φυσικό αέριο και για τον ηλεκτρισμό. Χρειαζόμαστε καλύτερα ευφυή ε, ηλεκτρικά δίκτυα και καλύτερη χρήση του άνθρακα. Στη Δανία Έχουμε τέτοιες μονάδες οι οποίες χρησιμοποιούν αυτό το 7%. Μπρετσίνα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η έκθεση αυτή επιτέλους συνετάχθη και θα ήθελα να συγχαρώ το συνάδελφο Μπούζεχ. Η αγορά αυτή όμως δεν είναι ανοιχτή στο τμήμα της Ευρώπης όπου ζω εγώ. Είναι μια ρυθμισμένη αγορά και δίνει προτίμηση στις ανανεώσιμες, κάτι το οποίο στρεβλώνει την αγορά. Η... Τα δίκτυα τα ηλεκτρικά μας δίκτυα δεν είναι επαρκή και τα ευφύ δίκτυα αποτελούν ακόμα θεωρία. Δεν έχουν εισαχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μία πλευρά της αγοράς υπόκειται σε μεγάλη στρέβλωση και δεν αποστέλουμε τα σωστά μηνύματα στους επενδυτές. Η τιμή της ενέργειας έχει καθήλωθεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να χτίσει μία παραδοσιακή μονάδα ενεργειακής απόδοσης. Χρησιμοποιούμε καφέ άνθρακα. Πολλοί θεωρούσαν το, τη χρήση φυσικού αερίου θα ήταν καλύτερη, αλλά δεν ισχύει αυτό πάντα. Εγώ μιλώ για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Δημοκρατία της Τσεχίας. Εδώ υπάρχει συνδεσιμότητα μεταξύ των τριών αυτών ε, χωρών. Υπάρχει μεγάλη επιδότηση που δεν χρειάζεται να οικοδομηθούν παραδοσιακές μονάδες. Δεν μπορούμε όμως να βασιστούμε μόνο σε ανανεώσιμες. Θα ήθελα μια γνήσια αγορά ενέργειας στην Ευρώπη και περισσότερη, μεγαλύτερη επικριτική στάση έναντι ημών όταν υποστηρίζουμε τις ανανεώσιμες. Δεν μπορούμε να προτρέχουμε δυστυχώς. Θα, πρώτα, θα πρέπει πρώτα να επιλύσουμε το θέμα των εφιών δικτύων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για ελεύθερο ανταγωνισμό έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν σταθερότητα, ασφάλεια και τις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Αυτό είναι ο απότερος στόχος και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που αντιτάσσεται στο άνοιγμα της αγοράς στην ενέργεια. Για να ανοίξουμε όμως την αγορά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για μια ελεύθερη και ανοιχτή αγορά. Μιλάμε για διασυνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η διασυνδεσιμότητα δεν ε, μπορεί παρά να προσκρούσει σε στενοπούς. Και στις βαλτικές χώρες δεν υπάρχει συνδεσιμότητα, διασυνδεσιμότητα. Οι μόνοι αγωγοί συνδέονται με τη Ρωσία, με την Gazprom που κατέχει το μονοπόλιο κατά 100%. Άρα δεν υπάρχει φυσική δυνατότητα να εισαχθεί ο ανταγωνισμός, όποια και να είναι τα νομοθετικά πακέτα. Ένα άλλο θέμα που εφήγει, δηλαδή οι ανανεώσιμες και οι επιδοτήσεις, θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι υπάρχει ένα διαφορετικό, σε κάθε χώρο υπάρχει διαφορετικό εθνικό σύστημα επιδοτήσεων και άλλο συσχετισμό επιδοτήσεων και όσο ανοίγει η αγορά αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει πραγματικό πρόβλημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι για να λειτουργήσει πραγματικά η αγορά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη για να υπάρχει διασυνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών μελών. Και έτσι μόνο θα μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά. Επίσης, χρειάζεται μία ενοποίηση στο σύστημα επιδοτήσεων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει πραγματικά να λειτουργήσει. Γιατί αν σε μία αγορά η, ο ηλεκτρισμός επιδοτείται κατά πολύ, τότε η άλλη χώρα βρίσκεται σε θέση μειονεξίας. Αυτό που θέλουμε είναι την καλύτερη τιμή για τον τελικό χρήστη και αυτός θα πρέπει να είναι ο απότερος στόχος. Χένιμ. Ευχαριστώ, πιστεύω ότι δεν τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν μας λένε ότι η αγορά δεν είναι ανοιχτή, ότι πρέπει να επελευθερώσουμε την αγορά, να είναι διαφανής και ούτω καθεξής, βασιζόμαστε σε αντικειμενικά δεδομένα. Ε, τομείς οι οποίοι έχουν δυσκολία προμήθειας, χώρες που έχουν δυσκολίες και θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι απελευθερώνοντας την αγορά θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ας δούμε ε, τι οδήγησε στην απελευθέρωση της αγοράς. Η αύξηση του ενεργειακού, κόστου, του ενεργειακού κόστους για τον καταναλωτή, για τις επιχειρήσεις και ακριβώς επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλούμε περισσότερο ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι παράγουμε, το οποίο σημαίνει ότι την μεταπολούμε. Και οι μικρές μονάδες που ανήκαν στα κράτη, σε εθνικές οντότητες, τώρα μεταπολούνται σε επιχειρήσεις. Άρα, στη δική μου περιφέρεια, μία μονάδα η οποία θα μπορούσε να παράγει ένα πλεόνασμα, κλείνει και η μεταπόληση δεν μπορεί να γίνει μεταπόληση σε άλλες χώρες. Θα σας πω τι θα γίνει στο τέλος. Θα έχουμε αύξηση του κόστους ενέργειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους φύλακες, διότι οι επιχειρήσεις δεν θα επενδύσουν εκεί που η αποδοτικότητα είναι χαμηλότερη και θα έχουμε μεγαλύτερο ευεργέτημα για τους μεγάλους ομίλους οι οποίοι κατέχουν και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Το λόγο έχει η Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση συνεχί. Ζούμε βέβαια στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και σας διαβεβαιώ πως σκοπεύουμε στην Κομισιόν να εφαρμόσουμε το σχέδιο δράσης και να προχωρήσουμε στο δυνατόν πιο γρήγορα στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για την ενέργεια μέχρι το 2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Συγητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευτυχώς στο τέλος της συζήτησης είχαμε και κάποια διαφωνία, οπότε αισθάνομαι κάπως καλύτερα. Αλλά χαίρομαι και το ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι υποστηρίζουν την ιδέα της εσωτερικής αγοράς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία είπατε. Θα ληφθούν υπόψη και θα είναι έτοιμοι βεβαίως τον επόμενο μήνα και πόσο θυμάμαι 20 Απριλίου νομίζω είναι οι προθεσμοί της τροπολογίας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες και η επόμενη συζήτηση του σχεδίου έκθεσης θα είναι τον Απρίλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ήμουν και σύντομος. Ευχαριστώ συναδελφέ Μπούζεκ και τώρα θα ζητήσω από τον Αλμπέρτο Ποτόσνικ που ε, διευθύνει το Άσερ να μας παρουσιάσει μια γνωμοδότηση που στενά συνδέεται με την έκθεση που μόλις μας παρουσίασε ο συνάδελφος Μπούζεκ. Το λόγο λοιπόν έχει ο Αλμπέρτο Ποτόσνικ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας σας όλα τα μέλη της Επιτροπής για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμεριστώ μαζί σας την άποψη της υπηρεσίας για τις ε, δυνατότητες, για τις δυνατότητες αγορών ε, εμείς ε, εξετάζουμε το πιθανό αντίκτυπο της μαζικής διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αναμένεται στα επόμενα χρόνια στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κατά πόσο το μοντέλο στόχων ηλεκτρισμού που είχε συμφωνηθεί πριν από κάποια χρόνια πρέπει να ανανεωθεί. Αυτά εν συντομία ε, περιλαμβάνονται στη γνωμοδότησή μας και αυτά αφορούν τον προβληματισμό μας σε αυτή τη φάση. Εξακολουθούμε να εκτιμούμε ωστόσο τον αντίκτυπο διαφόρων ε, ε, μηχανισμών αμοιβή στην εσωτερική αγορά ε, και τις δυνατότητες αυτών και γι' αυτό και θέλουμε να διατηρηθεί και να συνεχιστεί ο διάλογος για αυτό το θέμα μαζί σας. Όπως γνωρίζετε, στις 14 Νοεμβρίου ζητήσατε μια γνωμοδότηση από εμά για τις ε, αγορές ισχύω. Και τέσσερα συγκεκριμένα θέματα αναφέρονταν στην επιστολή σα και εδώ τα παραθέτω όχι με την ίδια σειρά, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελα να απαντήσω. Πρώτα, έχουμε μια αξιολόγηση των αναγκών επένδυσης για την ε, παραγωγή ε, μεταφορά και διανομή στα επόμενα δέκα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως τη δίσδυση των ε, ανανεώσιμων. Δεύτερη ερώτηση είναι το μέλλον της ενέργειας, της ενεργειακής αγοράς και πάλι υπό το φως της δίσδυσης των ανανεώσιμων πηγών και έπειτα το θέμα του ε, κατά πόσο απαιτείται η αναζήτηση αγορών ισχύως και ποιος είναι το, ποιο είναι το κατάλληλο γεωγραφικό εύρος και πώς θα υπάρξει διαβελιξία στις σχετικές αυτές αγορές αγορές και μιλάμε για τις βράχοι πρόθεσμες αγορές. Να μιλήσω για το πρώτο θέμα πρώτο και για εκτιμήσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, και οι Ευρωπαίοι φορείς, Ευρωπαϊκοί φορείς μάλλον, μετάδοσης ισχύω, μεταφοράς ισχύω. Οι επενδύσεις πάνω από 800 δις ευρώ θα χρειαστούν στον τομέα του ηλεκτρισμού. Τα 500 δε από αυτά δις θα αφορούν την παραγωγή ενέργειας. Και βέβαια η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, μάλλον παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα αντιστοιχεί στο 90% των νέων δυνατοτήτων. Το μείγμα λοιπόν παραγωγής το 20 θα είναι πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Και αυτό βέβαια α, επηρεάζει την μεταφορά και την Διανομή. Και 300 δις αναμένεται λοιπόν να χρειαστούν για επενδύσεις στη μεταφορά και στη διανομή, περίπου το 1 τρίτο αυτών στην μεταφορά και το 80% των νέων υποδομών θα συνδέονται με την ανάγκη ε, χρήσης των ανανεώσιμων. Αυτό συνδέεται και με τη διανομή, όπου σε κάποιο βαθμό πρέπει κανείς να στηρίξει την ανάπτυξη των ε, δεδομένων ε, ε, παραγωγών και διανομής. Επίσης θα χρειάζεται να συμμετέχει η διανομή και στην αγορά. Μια σημαντική πτυχή στην οποία θα ξανααναφερθώ. Να αναφερθώ τώρα σε τρεις ε, έννοιες που σχετίζονται με την ασφάλεια ανεφοδιασμού. Και αυτές είναι σημαντικές οι κατά τη γνώμη μας, όταν ε, πρέπει κανείς να δει την ε, σχέση ανάμεσα στην αγορά ενέργειας και τις, τις ρυθμίσεις περί ισχύως. Καταρχήν η παροχή, μάλλον η ασφάλεια ανεφοδιασμού, δηλαδή η δυνατότητα του συστήματος ηλεκτρισμού να παρέχει ηλεκτρισμό στους τελικούς χρήστες κάθετος πελάτες ε, σε με σταθερή ποιότητα και παροχή. Αυτό είναι ένας γενικός ορισμός. Τώρα πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένες έννοιες και διάφορες έννοιες εδώ μπορούν να εξεταστούν εάν εξετάσουμε τα διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Έχουμε δύο συγκεκριμένες έννοιες που έχουν σχέση με τους δικούς μας στόχους. Το πρώτο είναι η καταλληλότητα του πόρου, που είναι μια μακροχρόνια έννοια και αναφέρεται στη δυνατότητα ή στη διαθεσιμότητα επαρκών ικανοτήτων στο σύστημα ώστε να ανταποκρίνεται στη ζήτηση, ε, στη ζήτηση ανα πάσα στιγμή συμπεριλαμβανομένων και των σημείων εχμής. Ε, έπειτα υπάρχει η επιχειρησιακή αξιοπιστία που είναι ένας βραχυπρόθεσμος όρος και αφορά την διατήρηση της ευελιξίας του συστήματος ώστε να διατηρείται η ισορροπία ανα πάσα στιγμή και ιδιαίτερα σε σχέση με ε, ε, ξαφνικές αλλαγές στη ζήτηση ή μη, αναμενόμενες, μη αναμενόμενα προβλήματα στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Αυτό έχει να κάνει δηλαδή περισσότερο με την ποιότητα. Αυτά τα δύο θέματα έχουν διαφορετικό αντίκτυπο όσον αφορά την ικανότητα των αγορών να παρέχουν αυτές τις δυο Το μέλλον λοιπόν των ενεργειακών αγορών για ορθώς λειτουργούσα αγορά ενέργειας θα πρέπει να δίνει μηνύματα όσον αφορά την προώθηση της ασφάλειας ε, παροχής. Αυτό το πιστεύουμε κράδαντα. Γι' αυτό ο στόχος όσον αφορά την αγορά ενέργειας θα είναι να αρθούν οι υπάρχοντες φραγμοί. Στη συζήτηση που είχατε αμέσως πριν έγινε μια αναφορά στα, στους φραγμούς αυτούς οι κανόνες που αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουν στην τιμολόγηση, στο σχηματισμό της τιμής. Υπάρχουν ας πούμε ρητά ή ρητές ή άρρητες οροφές τιμών. Και πάλι υπάρχουν κανόνες της αγοράς αλλά και συγκεκριμένα μέσα. Πολύ περιορισμένη συμμετοχή δε της ζήτησης στις αγορές. Και η βασιζόμενη στην αγορά ζήτηση είναι σπάνια, ε, σπάνια μεταβλητή. Θα πρέπει να παραμείνει λοιπόν αυτό ως ε, βασική προτεραιότητα γιατί αποτελεί, δίνει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και, πρέπει, και είναι πιο ασφαλής βάση για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Ας περάσουμε τώρα στο πιο επίκαιρο πράγμα, δηλαδή το κατά πόσο χρειάζονται οι αγορές ε, είναι μια απλή ερώτηση, αλλά δεν έχει απλή απάντηση, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση σε σχέση με τα τελευταία 25 χρόνια. Και εξακολουθούν να γίνονται σχετικές συζητήσει. Η τρίτη οδηγία περί ηλεκτρισμού, που είναι τμήμα του τρίτου πακέτου, ε, συζητά τη δυνατότητα των κρατών μελών να εξασφαλίζουν ε, τις διαδικασίες ε, υποβολής τροπο, Υποβολή ε, προτάσεων για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί οι οποίοι εξετάζονται στα κράτη-μέλη. Δυστυχώ, αυτή τη στιγμή όλα αυτά γίνονται χωρίς κανένα συντονισμό και η εικόνα αυτή εδώ δείχνει την ισχύουσα κατάσταση όπως μπορέσαμε να συλλέξουμε τις σχετικές πληροφορίες, κυρίως από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, να δούμε ε, τους ε, μηχανισμούς ε, απόδοσης ανταμοιβή μάλλον της ισχύω. Οι χώρες που είναι σε κίτρινο είναι αυτές που εξετάζουν τη δυνατότητα εισαγωγής τέτοιων μηχανισμών. Οι πράσινες είναι αυτές που για την ώρα είναι μόνο αγορές ενέργειας. Να δούμε λοιπόν αν χρειαζόμαστε αγορές ισχύω. Καταρχήν, μια αγορά ενέργειας θα μπορούσε να δώσει επάρκεια και επάρκεια, καταλληλότητα μάλλον πόρων και ευελιξία του συστήματος. Το θέμα είναι κατά πόσο η αγορά λειτουργεί χωρίς ε, εμπόδια. Δηλαδή μπορεί να ανταποκριθεί στα μηνύματα των τιμών και τα μηνύματα αυτών των τιμών θα πρέπει να μπορούν να κυμαίνονται ελεύθερα και να αντικατοπτρίζουν την σχέση μεταξύ ζήτηση και παροχής. Σε τιμές δηλαδή όπου είναι λιγοστή ενέργεια θα πρέπει οι τιμές να μπορούν να αυξηθούν στο επίπεδο του κόστους. δεν έχουμε ε, έτσι πρόβλημα με την ασφάλεια ανεφοδιασμού, τουλάχιστον όσον αφορά την καταλληλότητα. Έχουμε επίσης άλλες προϋποθέσεις και όρους που θα πρέπει να πληρούνται, έτσι ώστε οι αγορές ενέργειας να εξασφαλίζουν την ασφάλεια ανεφοδιασμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι, έχουν, ότι υπάρχουν σταθερά πολιτικά καθεστώτα, καθώς και ότι οι, οι πολιτικοί θύνοντες θα αντισταθούν στον πειρασμό να παρεύουν όταν αυξάνονται οι τιμές και παραμένουν σε ψηλά επίπεδα. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν την απόδοση των επενδύσεών τους σε σχετικά τακτικές αλλαγές, σχετικά αλλα... Ε, τακτικές αλλαγές τιμών. Μέχρι ότου λοιπόν να πληρούνται αυτές, αυτοί οι όροι δεν υπάρχει εγγύηση ότι μια αγορά αποκλειστικά ενέργειας θα μπορεί να δώσει την ε, καταλληλότητα των πόρων αλλά και την επαρκή ευελιξία. Ακόμα και αν αρθούν όλα τα εμπόδια και υπάρχει ολοκληρωμένη αγορά. Μπορεί λοιπόν μέχρι τότε να χρειαζόμαστε, μέχρι ότου δηλαδή πληρούνται αυτοί οι όροι και γι' αυτό και προσπαθούμε να αφαιρέσουμε τις τρευλώσεις και τα εμπόδια στην αγορά. Πιστεύω λοιπόν πως μέχρι τότε ίσως να χρειάζεται να συμπληρώσουμε την ενεργειακή αγορά με με ε, πρόσθετες ρυθμίσεις ε, και χρησιμοποίησα τη λέξη ρυθμίσεις επίτηδες. Θα σας πω γιατί σε λίγο. Στόχο θα πρέπει να έχουν να προωθούν την καταλληλότητα και την ευελιξία. Και εν πάση περιπτώσει μια ορθώς λειτουργούσα ενεργειακή αγορά δίνει καλύτερο χώρο για αυτές τις επιπλέον ρυθμίσεις και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται η πρόοδος και η αναζήτηση τη ασφάλεια ανεφοδιασμού να μην εμποδίζει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Αυτέ οι επιπλέον ρυθμίσει που μπορεί να ληφθούν υπόψη δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν, να στρεβλώνουν τη λειτουργία της αγοράς ε, ενέργειας και ιδανικά να ε, την επηρεάζουν μόνο σε βαθμό που η ενεργειακή αγορά δεν θα αποδίδει και θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ουδέτερε στις υπόλοιπες ε, φάσεις. Όσον αφορά τώρα το γεωγραφικό φάσμα, οποιασδήποτε ρύθμιση περί αμοιβή ισχύω, για την ισχύ μάλλον, αυτό εξαρτάται από τις διάφορες δικαιοδοσίες που θα πρέπει να αποφασίσουν ή να ορίσουν την τις κοινέ προδιαγραφές καταλληλότητας και ασφάλειας. Και αυτό δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο σε ένα πλαίσιο εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού. με η στρέβλωση στην εσωτερική αγορά θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί εάν ε, μπορούσαν να συμμετέχουν τα γειτονικά κράτη στην ε, αγορά και αυτό να το διευκρινίσω γιατί κάποιες φορές αυτό προκαλεί ανησυχία. Η συμμετοχή στους πόρους που το είναι τοποθετημένοι σε άλλα κρατημέλη, τουλάχιστον όσον αφορά την καταλληλότητα, δεν απαιτεί την ε, μείωση της ισχύω που ξέρουμε πως καλύτερα χρησιμοποιείται για εμπορικές συναλλαγές. Αλλά σε αυτό να μπορέσουμε να επανέλθουμε αργότερα. Γι' αυτό λοιπόν η εισαγωγή εθνικών μηχανισμών θα πρέπει να συνοδευτεί από μια στιβαρή μελέτη αντικτύπων που θα λαμβάνει υπόψη τα συνοριακά φαινόμενα και επίσης πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει κάποια προσδοκία πως οι μηχανισμοί αυτοί θα παραμείνουν επάπειρον. Γιατί έτσι όπως ε, βελτιώνονται οι αγορές ε, ενέργειας μπορεί να χρειαστεί να τα επανεξετάσουμε και η υπηρεσία μας παραδείγματο χάρη αυτή τη στιγμή κάνει μια αξιολόγηση ε, του αντικτύπου των διαφόρων μηχανισμών. Οπότε στο μέλλον μπορεί να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το ζήτημα. Οπότε, η συμβατότητα τη συμβατότητα οποιασδήποτε αμοιβή θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Να έρθω τώρα στην ευελιξία. Και η ευελιξία λοιπόν πρέπει να προωθηθεί από τα βραχυπρόθεσμα μηνύματα των τιμών. Αυτή τη στιγμή έχει διαφαλιστεί η επάρκεια. Πρέπει τότε να δοθούν τα κατάλληλα μηνύματα για ευελιξία από τις βραχυπρόθεσμες αγορές και στο πλαίσιο αυτό της λειτουργίας των συστημάτων και της εξορρόψης έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τις διασυνοριακές αγορές για να είναι σαφέστερα τα μηνύματα της ε, ανεπάρκειας και να προωθηθούν οι επενδύσεις σε νέες ε, ευέλικτες δυνατότητες ε, παραγωγής για να υπάρξει καλύτερη δυνατότητα μεταξύ των διαχειριστών του δικτύου για την ε, καταμέτρηση, την ανταλλαγή και τον διαμοιρασμό τέτοιων προϊόντων εξορόψης και βέβαια για να διευκολυνθεί η συμμετοχή στις αγορές αυτές. Και βέβαια πρέπει να ενισχύσουμε και τις ε, νέες ε, τεχνολογίες, ειδικά στις αγορές συμπληρωματικών υπηρεσιών. Για να καταλήξουμε λοιπόν όσο οι αγορές ενέργειας δεν επιτρέπεται να λειτουργούν ε, ανεμπόδιστες, δεν υπάρχει εγγύηση πώς θα μπορέσουν από μόνες τους να δώσουν το απαραίτητο επίπεδο επάρκειας ε, και ευελιξίας του συστήματος. Οπότε η βασική μας προσπάθεια θα πρέπει να είναι στο να αφαιρέσουμε τα εμπόδια και να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά η ασφάλεια της παροχής του ή εξυπηρετείται καλύτερα από το να λειτουργεί επαρκώς η αγορά και με το να δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η πλήρη συμβατότητα οποιοδήποτε εθνικού σχεδίου θα πρέπει να διασφαλιστεί συμβατότητα με την εσωτερική αγορά ενέργειας και βεβαίως ένα σωστό κλίμα για τις επενδύσεις θα προωθήσει τη συμμετοχή νέων τεχνολογιών και θα αυξηθεί έτσι η ζήτηση ε, των ε, συμπληρωματικών υπηρεσιών. Αυτά εν ολίγης περιέχονται στη γνωμοδότησή μας, όπως είπα ακόμα είναι υπό σύνταξη και καλωσορίζουμε την ευκαιρία να ε, δούμε τα μελλοντικά αποτελέσματα μαζί σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δώσατε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ποτότσνικ. Εμείς ως Επιτροπή είχαμε ζητήσει ε, από την υπηρεσία σας να κάνει αυτή τη μελέτη. Τον λόγο έχει προφανώς ο συνάδελφος ο κύριος Μπουζέκ. Uh, um, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη στην εσωτερική μας αγορά τις δυνατότητες και με ποιο τρόπο αυτές μπορούν να επηρεάσουν την εσωτερική αγορά ενέργειας. Αν είναι οι αγορές κλεισμένες και διαχωρισμένες και εθνικές, τότε η οικοδόμηση τέτοιων δυνατοτήτων ε, μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και περισσότερους διαχωρισμούς, γιατί δεν είμαστε ανοιχτοί ε, εκτός του κράτους μέλους ο καθένας. Στην περίπτωση των διασυνδέσεων και στην περίπτωση που λειτουργεί η εσωτερική αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε η οικοδόμηση περαιτέρω δυνατοτήτων να στηρίξει την αγορά και να μας δώσει μια πραγματική ασφάλεια παροχής ενέργειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε να επαναλάβουμε το εξή. Το σημαντικότερο για εμάς είναι η ε, επένδυση στις υποδομές. Χρειαζόμαστε 140 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρόσεχες μέλλον και από την άλλη πρέπει να δημιουργηθεί, όπω είπα, αυτή η δυνατότητα παραγωγή Γιατί χρειαζόμαστε συνολικά ένα 3 εκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2020, αν είναι να έχουμε πραγματική επάρκεια και να πάει η οικονομία μας προς λιγότερες εκπομπές και να υπάρξει δυνατότητα να ε, μειωθούν οι τιμές. Ποτέ δεν θα είναι χαμηλές στο μέλλον. Αλλά να μειωθούν και γι' αυτό χρειάζεται, όπως είπα, περισσότερη ε, δυνατότητα παραγωγής και να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Οπότε θεωρώ πως η πραγματική αφετηρία σε οποιαδήποτε συζήτηση είναι η διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών και ε, μια πραγματική ενιαία αγορά για την ενέργεια. Ευχαριστώ. Κορέα Ντεκάμπος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ποτότσνικ για την εξαιρετική του παρουσίαση. Εμείς γνωριζόμαστε από όταν είχαμε συνεργαστεί στα ενεργειακά δίκτυα και βεβαίως έχουμε πάρα πολλά κοινά. Να ξεκινήσω συγχαίροντας σας για την μεθοδολογία της ε, παρουσίασής σας. Ε, Εξετάζετε τη ζήτηση αντί για την προσφορά. Στο παρελθόν κοιτάγαμε την προσφορά και προσπαθούσαμε να εναρμονίσουμε την προσφορά. Τώρα επιτέλους αντιστρέφεται αυτή η τάση. Κοιτάμε τις μελλοντικέ ανάγκες και δεν κοιτά μόνο τι θα κάνουμε την ε, ε, παραγωγή. Δεύτερον, χαίρομαι για το ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην επιχειρησιακή αξιοπιστία όταν μιλάμε για την ασφάλεια της ε, παροχής και χαίρομαι για το ότι δέχεστε αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε στην νομοθεσία όσον αφορά τον ε, συντονισμό χωρίς αποτελεσματικό επιχειρησιακό συντονισμό θα έχουμε αποτυχίες στον ε, τομέα της ασφάλειας παροχής ενέργειας. Ε, το τρίτο αφορά τις τιμές και το μηχανισμό στο εθνικό επίπεδο για να ρυθμιστούν οι τιμές. Πάντα οι πολιτικοί έχουν δύσκολες σχέσεις ε, με τις ρυθμιστικές αρχές γιατί τα κράτη-μέλη θέλουν να μην επιτρέπουν στις τιμές να αυξηθούν ή να επιβάλλουν πλαφών, τέτοια πράγματα κάνουν. Και ε, κάποια φορά αυτό είναι ε, στρέβλωση του ανταγωνισμού. Βεβαίως ε, πρέπει να αντιληφθούμε πως το κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του πολιτική λογική. Και σε καιρούς κρίσιμους είναι δύσκολο να ε, επιτραπεί η άνοδος των τιμών του ηλεκτρισμού. αλλά έχουμε έναν ξεκάθαρο διάλογο και καλύτερη σχέση μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και κρατών μελών. Και εδώ πέρα συμφωνώ μαζί σας, ε, οι ανοιχτές ε, αγορές και τα μηνύματα μέσω των τιμών είναι κάτι τόσο σημαντικό. Τέλος, έχω κάποιες αμφιβολίες. Ε, η αγορά αυτή δεν είναι τέλεια. πρέπει να έχουν ε, οι ρυθμιστικές αρχές την δυνατότητα να αποτρέψουν τις άσχημες επιπτώσεις στους ε, καταναλωτές. Το βλέπουμε ελάχιστα από την πλευρά του καταναλωτή. Πρέπει λοιπόν και η ειδική υπηρεσία και όλες οι ρυθμιστικές υπηρεσίες ε, πρέπει να θεωρούν αυτούς όχι μόνο ρυθμιστές της αγοράς, αλλά κυρίως ως πρόσωπο ε, του καταναλωτή που χρειάζεται καλύτερες τιμές. Τελευταία ερώτηση. Εάν ο ανταγωνισμός είναι το καλύτερο περιβάλλον για την καινοτομία. Αυτό είναι ένα σωστό ερώτημα. Ίσως ναι, ίσως όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρόντι έχει το λόγο ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Ποτότσνικ για την ε, εισήγησή του. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναστρέψουμε αυτή τη λογική, διότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε ένα πέρασμα από, τα, από τις ορυκτές πηγές ενέργειας, τις ανανεώσιμες. Να δούμε και την αιωλική ενέργεια καθώς και τη φωτοβολταϊκή. Θα πρέπει να υπάρχει να χρησιμοποιηθούν προγενέστερα πριν από οτιδήποτε άλλο και θα πρέπει να δούμε τη σωστή διάσταση του ηλεκτρικού δικτύου που δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊκής ε, εμβέλειας αλλά που παράλληλα θα πρέπει να έχει χαμηλό, ε, χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον αν λάβουμε υπόψη τη χρήση των ηλεκτρικών δικτύων και θα πρέπει να δούμε την ευρωπαϊκή διάσταση των δικτύων πρωτίστως. Αυτό είναι ένα προγενέστερο σχήμα εάν θέλουμε πραγματικά να εκμεταλλευτούμε τις ανανεώσιμες διότι με το ευρωπαϊκό δίκτυο θα μπορούσαμε να έχουμε ευρία χρήση της αιωλικής και να χρησιμοποιήσουμε και την υδροηλεκτρική ενέργεια, κάτι το οποίο γίνεται και μέχρι τούδε. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τα υδροηλεκτρικά φράγματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως στήριξη της αιωλικής με σχήματα τα οποία να είναι προβλέψιμα. Έχουμε λοιπόν μία επιλογή ενώπιόν μας. Ιδιαίτερα ως προς τις επενδύσεις των ηλεκτρικών δικτύων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι, θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκής εμβέλειας. Διαφορετικά δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Ε, τα υδροηλεκτρικά φράγματα μπορούν να οδηγήσουν σε άμεση επέμβαση χρησιμοποιώντας και έναν ε, σύμικτο συμπληρωματικό ε, κύκλο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι και το επιπρόσθετο κόστος του άνθρακα. Και γι' αυτό χρειάζεται διαχείριση ενός ε, ηλεκτρικού δικτύου που πρέπει οπωσδήποτε να είναι ευρωπαϊκής εμβέλειας. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτή την εξέλιξη του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας. Γιατί θα πρέπει να, κατανοήσουμε ότι τα κράτη-μέλη από μόνα τους δεν μπορούν να εγγυηθούν στους καταναλωτές ε, τη δυνατότητα προμήθειας ενέργειας καθώς και την τήρηση των προδιαγραφών προς το περιβάλλον Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω ήθελα να πω στον Αλμπέρτο πως χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και ακούω τα όσα έχεις να μας πεις και οι συνάδελφοι να με συγχωρήσουν για να σας, γιατί θα σας θυμίσω πως ήμουν εισηγητής για το ΑΣΕΡ το τελευταίο περασμένη θητεία και γι' αυτό και συνεχίζω να ενδιαφέρομαι για τις δραστηριότητες και την επιτυχία σας. Μέσα στην εντολή συμπεριλαμβανόταν ε, και το... η σημερινή σας παρουσίαση, ε, δηλαδή ότι θα έπρεπε να έρχεστε στο Κοινοβούλιο τακτικά και να μας χρησιμοποιείτε ως μια ε, βάση για να δώσετε κωδικοποιημένα μηνύματα για το πού θέλετε να πάτε και τι θέλετε να κάνετε προς την Κομισιόν. Μήπως κάτι τέτοιο θέλετε να μας πείτε όταν λέτε ότι οι αγορές δεν λειτουργούν απόλυτα ελαστικά και καταλή. Τέλο, Να ρωτήσω λοιπόν την πρώτη μου ερώτηση, Πρόεδρε. Σε ποιο βαθμό μπορεί η υπηρεσία να καλύψει οποιασδήποτε νομικές, νομικά ελλείμματα για την προώθηση και την εξασφάλιση της, του πλήρους ανταγωνισμού στις αγορές. Είχαμε αυτή την πρόθεση ότι δηλαδή θα μπορούσατε με τη μεγαλύτερη ευελιξία που έχει μια αριθμιστική τέτοια υπηρεσία να το κάνει αυτό. Μπορείτε αυτό να το σχολιάσετε. Αν δεν είστε σε θέση να λύσετε όλα τα προβλήματα και δεν αναμένω να είστε σε θέση να τα αντιμετωπίσετε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω, εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε, γιατί εσείς αναφέρατε διάφορα προβλήματα, ελλείψεις, ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Ο Επίτροπος χθε το βράδυ έλεγε ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η οικονομική κατάσταση σε 12 μήνες, τι να λέμε για 5 χρόνια ή 10 χρόνια. Εσείς λοιπόν και οι διαχειριστές του δικτύου καλείστε να αντιμετωπίσετε επιτόπου την κατάσταση. Και τελευταία μου παρατήρηση, Πρόεδρε μετά από τα όσα άκουσα και χτες το βράδυ, ήταν αυτή η πρόκληση στο οικονομικό περιβάλλον να βρούμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε για να επενδύσουμε στις παραγωγικές δυνατότητες, τη διανομή και τη, μετα... τη μεταφορά και τη διανομή της ισχύω που χρειαζόμαστε. Και ο Πέτροπος είπε, παρατήρησε πως ο κόσμος δεν έχει καμιά όρεξη να επενδύσει. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάτι, να προτείνουμε κάτι για να διευκολύνουμε τις κεφαλαγορές και να τις καθοδηγήσουμε σε πολύ λογικές κατά τη γνώμη μου μακροχρόνιες επενδύσεις με καλή απόδοση. Τι μπορείτε να προτείνετε. Ευχαριστώ. Ο Μπαλτσούτης, παρακαλώ. Ευχαριστώ yra pateikta ir, šitas klausimas tikrai Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η παρουσίαση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Τσίτσεστερ για την παρέμβασή του. Χτες είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Επίτροπο τον κύριο Έτιγκερ για το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θεωρώ πως ε, και για το μέλλον ε, πρέπει να θέσουμε στόχους ε, μεταξύ των οποίων στόχων πρέπει να είναι και οι τιμές της ενέργειας. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Οι τιμές της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και πρέπει να μειωθούν. Και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, γιατί αφορά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η οποία κινείται μέσα στις παγκόσμιες ε, αγορές. Εσείς μιλήσατε βεβαίω πω κάτι τέτοιο θα αποτελέσει στρέβλωση των αγορών. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου οι συμφωνίες αυτές. Ε, ε, δεν θα είναι ε, υποχρεωτικές. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν και να αποτρέψουν τις διακυμάνσεις των τιμών, γιατί σε κάποιες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο οι τιμές. Γι' αυτό έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Το εάν δηλαδή οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές για τα δίκτυα και οι κώδικες για τα δίκτυα θα έχουν εγκριθεί ως το 2014. Επίσης τίθεται ένα άλλο ερώτημα όσον αφορά τον συντονισμό των περιφερειακών πρωτοβουλειών και την ανάγκη των απαραίτητων ε, υποδομών. Εξίσου σημαντικά ερωτήματα όπως και οι δραστηριότητες των ρυθμιστικών αρχών για τη ρύθμιση των ε, τιμών. Γιατί αυτή τη στιγμή οι αρχές αυτές ε, παίζουν και θετικό και αρνητικό ρόλο. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Ποτότσνικ ε, για την παρουσίασή του, αλλά πρέπει να πω πως ε, την βρήκα κάπως ακαδημαϊκή και θεωρητική και αναρωτιέμαι ποιες είναι οι άμεσες ε, επιπτώσεις της για τη Γερμανία καθώς προσπαθεί να αντικαταστήσει τα πυρηνικά εργοστάσια με λιγνητικά ή το τι σημαίνει για τη χώρα μου καθώς αντιμετωπίζουμε έναν γκρεμό πλέον παραγωγικής δυνατότητας. Ε, κλείνουμε τα πυρηνικά εργοστάσια και τα εργοστάσια άνθρακα και δεν ξέρουμε με τι θα τα αντικαταστήσουμε. Κύριε Ποτότσνικ, με εξέπληξαν τα νούμερα που παρουσιάσατε και αναρωτιέμαι αν ε, θα μας δώσετε αντίγραφα της παρουσίασής σας, γιατί θα τα ήθελα. Αλλά ε, ξεκαθαρίστε μου το εξής. Ε, έχω την εντύπωση, πως είπατε, πως θα χρειαστούμε 300 δισεκατομμύρια ευρώ για δίκτυα διανομής και 80% από αυτά αφορούν το ζήτημα της αντιμετώπισης των ανανεώσιμων. Τεράστια ποσά. Δεύτερον, συζητήσαμε ξανά τις σχετικές πληρωμές ε, που πάλι ε, ε, σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των ανανεώσιμων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως οι πληρωμές αυτές των δυνατοτήτων είναι απλά μέτρο της αναποτελεσματικότητας γιατί χρειάζεται ένα backup πάντα για να, μια εφεδρεία για να στηριχθούν οι ανανεώσιμες και είχαμε μια συζήτηση πρόσφατα και ακούστηκαν πάρα πολλά ε, νούμερα για την ανταγωνιστικότητα των φωτοβολταϊκών και μιλήσανε για ισότητα στο δίκτυο. Αλλά όταν μιλάνε για το, κόστο των, κόστος των ανανεώσιμων, η παραγωγή σχετική, μιλάνε μόνο για το κόστος της ενέργειας που παράγουν. Οπωσδήποτε, όμως θα πρέπει να προσθέσουν και το τεράστιο κόστος προσαρμογής του δικτύου. Και των λοιπόν δυνατοτήτων χωρίς τα οποία δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες και άρα είναι πολύ πιο ακριβές από τα, πολύ, πολύ πιο ακριβές από τα νούμερα που κυκλοφορούν συνήθως. Επίσης μου πρόξενε η εντύπωση το ότι δημιουργείται ένα σύστημα με πάρα πολλές μεταβλητές. Και ως ε, πρώην μαθηματικός αναγνωρίζω πως είναι ένα περίπλοκο ή και χαοτικό σύστημα. Και ως πρώην μαθηματικός σας λέω πως ένα από τα μεγάλα χαρακτηριστικά των χαοτικών συστημάτων είναι πως τα αποτελέσματα διαφέρουν πάρα πολύ με πολύ μικρές αλλαγές στις αρχικές συνθήκες και άρα τέτοια συστήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθούν όσον αφορά τα αποτελέσματα και τη συμπεριφορά τους και υποψιάζομαι πως τα αποτελέσματα από το σύστημα που δημιουργείται θα είναι διαφορετικά από τις προσδοκίες σας όπως ακριβώς και διαφορετικά ήταν τα αποτελέσματα του συστήματος εμπορίας εκπομπών από τις προσδοκίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να θυμίσω στον συνάδελφο Χέλμερ καθώς και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, ότι στάλει εχθές η έκθεση μέσω mail. Θα το βρείτε λοιπόν στα mail σας την παρουσίαση του κυρίου και η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. είναι σημαντικό το να ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας και να δημιουργήσουμε και δίκτυα ή πλέγματα με αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να πούμε ε, ότι θα πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, γιατί όταν προετοιμάζουμε μια έκθεση στην Επιτροπή Ρέτζι ακριβώς ε, για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον αντίκτυπό του στην ενέργεια, ε, δώσαμε λίγα, προβλέψαμε λίγα κονδύλια για τις υποδομές για το φυσικό αέριο που είναι μια σημαντική ενέργεια για την συμπαραγωγή ε, και γι' αυτό και τώρα είμαστε σε δύσκολες διαπραγματεύσεις έτσι ώστε από τη μια πλευρά να, έχουμε, ε, να καλύψουμε τη χρηματοδότηση αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτό να γίνει με τα κονδύλια που στόχο έχουν την περιφερειακή ανάπτυξη. Εγώ παρακολουθούσα τη συζήτηση για το άνοιγμα των αγορών ισχύω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμής στο έγγραφό της σε σχέση με την λειτουργία των αγορών ενέργειας ε, είπε ε, πως τελικά μπορεί να δώσουν αρνητικά αποτελέσματα ή λανθασμένα αποτελέσματα οι αγορές ισχύω σε σχέση με τις τιμές. Άρα λοιπόν η ερώτησή μου είναι μήπως είναι ανεπαρκές ανεπαρκέ, ε, οι προτάσεις της Κομισιόν, μήπως τα, τα όσα προτείνετε πιστεύετε πως θα καλύψουν αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Έχω μια ερωτησούλα μόνο. Έχουμε το μείγμα ενέργειας για τις χώρες και έχουμε κάποιες γενικές πολιτικές. Αλλά πώς μπορούμε να εμποδίσουμε λόγω αυτής της ε, ε, μη σταθερής ροής ανανεώσιμης ενέργειας να κόβουμε ε, η χρήση του φυσικού αερίου που είναι το, η ενέργεια που μολύνει λιγότερο το περιβάλλον ενώ αυξάνεται η κατανάλωση άνθρακα. Θα πρέπει να καλύψουμε, να, να σκεφτούμε περισσότερο γιατί είναι ίσως εύκολο, πιο εύκολο να κλείνει κανείς τον γκάζι από ότι να πάβει να χρησιμοποιεί τον άνθρακα. Αυτή είναι μια ίσως τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση. Ή μήπως κρύβεται πίσω από εδώ κάτι. Δηλαδή υπάρχουν ε, ε, συγκαλυμμένα προβλήματα όσον αφορά τη ρήπανση και τις ε, επενδύσεις. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνονται έτσι οι παρεμβάσεις και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ποτόσνικ για να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα, αλλά να ζητήσω εξ αρχής συγγνώμη αν τυχόν κάτι ξεχάσω αν και τα έχω σημειώσει όλα. Επίση, θέλω να καταστήσω σαφέ όπω φαντάζεστε. Θα σας πω εξ αρχή ότι ισχύουν διαφορετικά πράγματα στα κράτη-μέλη και απόψεις και μεταξύ των ε, ρυθμιστών σε σχέση με τις αγορές ισχύω. Ε, κάποιες φορές θα σας δώσω τη δική μου προσωπική άποψη Αν και θα προσπαθήσω να μείνω στα όσα πιστεύω πως θα στήριζε η κοινότητα των ρυθμιστών στην Ευρώπη. Για τον κύριο Μπούζεκ, ελπίζω το μήνυμά μου να ήταν ξεκάθαρο. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας Ηλεκτρική ενέργεια πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα για δύο λόγους, τουλάχιστον δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι η πιο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπο για να ανταποκριθούμε στη ζήτηση και γιατί σε κάθε περίπτωση είναι η καλύτερη βάση για οποιαδήποτε επιπλέον ρύθμιση, εάν χρειαστεί επιπλέον ρύθμιση. Νομίζω ότι από αυτού είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο και θα πρέπει να πω ότι έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες, όχι μόνο για να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το νέο σύνολο κανόνων μέσω των κατευθυντηρίων γραμμών αλλά και του κώδικα που έχουν φτιάξει οι χειριστές μεταφοράς συστημάτων μεταφοράς αλλά και επίσης γιατί η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει συνολικά. Η ζήτηση είναι σημαντική και ο κύριος Κορέντε Κάμπος το τόνισε αυτό. Μάλιστα, όταν πρόκειται για η επιχειρησιακή αξιοπιστία, η ζήτηση είναι ο φθηνότερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Και με τη μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων και με με αυτή την ε, μεταβλητή των ανανεώσιμων, την ε, διακύμαση των ανανεώσιμων, όπως θα μπορούσαμε να την πούμε, μπορούμε κάποιες φορές βέβαια αφισβητείτε το πόσο διακύμανση ε, υπάρχει, πόση διακύμανση υπάρχει. Με πάση περιπτώσει, η επιχειρησιακή αξιοπιστία είναι θέμα και η ζήτηση είναι πολύ σημαντική το κόστος τώρα βέβαια οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν στο δυνατό πιο προσιτές Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε συνολικά είναι να μειώσουμε το συνολικό κόστος παροχής και ασφάλειας εφοδιασμό. Δεν είναι μόνο η τιμή στην αγορά ενέργειας που μετρά, αλλά και όλα τα άλλα κόστη που εμπλέκονται. Αν συγκρίνουμε τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας χωρίς κανένα φραγμό μια ορθώς λειτουργούσας της αγοράς ενέργειας με τη διανομή όπου υπάρχουν ε, οροφές στις τιμές κτλ, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πλήρες κόστος. Κύριε Πρόντιν, ελπίζω να μπορώ να σας καθησυχάσω για το ότι Υπάρχει, γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την επάκταση του δικτύου. Και μετά από το τρίτο πακέτο, πριν από δύο-τρία χρόνια, τα σχέδια ανάπτυξης δικτύου ε, αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο για τον ηλεκτρισμό όσο και για το φυσικό αέριο. Είναι δεκαετές το πρόγραμμα ανάπτυξης ε, και το σημείο αναφοράς είναι το σχέδιο των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ε, για την επέκταση του πλέγματος. Το πακέτο υποδομών που θα υιοθετηθεί σύντομα επίσης θα τονίσει τα σχέδια κοινού, κοινής ωφέλειας, που είναι αυτά τα οποία ε, καλύπτουν πάνω από ένα κράτος μέλος, Δίνεται δηλαδή περιφερειακή έμφαση στην ανάπτυξη των δικτύων και σαφώς ευρωπαϊκή διάσταση στον σχεδιασμό των δικτύων. Ελπίζω πως αυτό λοιπόν θα καθησυχάσει τις δικές σας ανησυχίες. Για τον κύριο Τσίτσεστερ, δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ κώδικες αλλά κάποια μηνύματα ε, θα έπρεπε να προκύψουν σαφώς από την γνωμοδότηση και την παρουσίασή μου. Οι φραγμοί πρέπει να έρθουν για την ορθή λειτουργία της αγοράς ενέργειας για πολλούς λόγους, όχι μόνο για να εξασφαλίσουμε την καταλληλότητα και την αξιοπιστία. Ως υπηρεσία δεν έχουμε αρμοδιότητα να παρέμβουμε άμεσα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά. Είμαστε τμήμα της διαδικασίας σχεδιασμού των κανόνων, παρακολουθούμε τις αγορές και μάλιστα πιθανότατα η βασική μας συμβολή, η πιο πολύτιμη συμβολή μας αυτή τη στιγμή είναι οι γνωμοδοτήσεις που μπορούμε να δώσουμε ή να ζητήσουμε και η δραστηριότητα παρακολούθησης και παρουσιάσαμε τον περασμένο Νοέμβριο την πρώτη μας έκθεση ε, για την αγορά όπου εντοπίσαμε φραγμούς, τάσεις στις ωραίες ενέργειες και φέτος η έκθεσή μας θα αναφέρεται συγκεκριμένα στους φραγμούς για την ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας. Αυτή είναι η συμβολή μας λοιπόν για την ώρα και ελπίζουμε και άλλα, άλλοι θεσμοί που έχουν ε, αρμοδιότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα σημειώνουν τα πορίσματά μας και θα ενεργούν αντιστοίχως. Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη ανέφερα, καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια από τότε που φτιάχτηκε η υπηρεσία μας πριν από δύο χρόνια για να προωθήσουμε την εφαρμογή των κανόνων όταν έχουν υιοθετηθεί και ακόμα και πριν να υιοθετηθούν, γιατί διαφορετικά είναι απίθανον να επιτύχουμε την ημερομηνία στόχο του 2014. Τώρα, όσον αφορά την ελκυστικότητα του τομέα ενέργειας για τα κεφάλαια, δεν είμαι επενδυτή ούτε τράπεζα, επενδυτική τράπεζα που δεν μπορώ να απαντήσω άμεσα λοιπόν, αλλά από πλευρά μα αυτό που θα μπορούσαμε να προτείνουμε ένα σταθερό ρυθμιστικό και ε, πλαίσιο πολιτικής. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε το ρυθμιστικό κίνδυνο που είναι ένα κίνδυνο που δεν αρέσει καθόλου στις αγορέ, γιατί πολύ δύσκολα μπορούν να τον ξεπεράσουν ή να τον προβλέψουν. Από τη δική μας πλευρά λοιπόν αυτή είναι η πρόκληση και γι' αυτό και πιέζουμε για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς γιατί αυτό θα είναι ε, μια επιτυχία που θα είναι η καλύτερη εγγύηση για σταθερό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Τώρα, υπάρχουν διάφορα προγράμματα στήριξης στις διάφορες αγορές, υπάρχουν διάφοροι κανόνες που ισχύουν στις διάφορες αγορές. Τώρα, η ολοκλήρωση των αγορών θα πρέπει να επιτρέψει και την σύγκληση του τιμών. Πλήρη σύγκληση τιμών βέβαια δεν μπορεί να είναι ο στόχος. Μπορεί να έχουμε κάποια απόκληση αν το κόστος της πλήρους ε, σύγκλησης τιμών είναι υπερβολικό. Αλλά για να δώσουμε ένα παράδειγμα θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά απλά βελτιώνοντας τους κανόνες Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι επήλθε μια συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ολλανδίας και ε, είδαμε ότι η σύγκληση τιμών ε, ανήλθε από 12%, από 12 σε 78%. Και συνεπώς ε, βελτιώσαμε τους κανόνες. Δεν, έγινε, δεν έγιναν επενδύσεις στις υποδομές. Μιλήσαμε λοιπόν για σύνδεση αγορών στη συγκεκριμένη περίπτωση και όχι έργα υποδομής. Προσπαθήσουμε λοιπόν, τα, προωθούμε λοιπόν τις κατευθυντήριες γραμμές για τα δίκτυα μέχρι το 13. Μέσα στο 13 θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για τις ανανεώσιμες όλες τις δαπάνες. Μιλάμε για 300 δις για τη διαβίβαση και το 80% των υποδομών θα καλυφθεί από τα 100 δις. Αυτό σχετίζεται με τις ανανεώσιμες. Οι ανανεώσιμες αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ανάπτυξη δικτύων. Υπάρχει μία αλλαγή. Το μέλλον των δικτύων ηλεκτρισμού, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα έχει την ίδια εικόνα που είχαμε μέχρι του παρόντος. Τέλος, και ελπίζω να μην ε, ε, άφησα ανοιχτά πεδία, τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκα αφορούν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Μιλάμε και για επενδύσεις βεβαίως, ε, για δίκτυα φυσικού αερίου. Εδώ υπάρχει μία διαφοροποίηση, διότι εδώ υπάρχει άμεση συνδεσιμότητα με τις ανανεώσιμες. Το φυσικό αέριο θα πληγεί περισσότερο από τις ανανεώσιμες. Πρώτον, διότι ήδη υπάρχει ο μεγάλος ανταγωνισμός των ανανεώσιμων ως προς τις μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου, πολύ περισσότερο, αλλά το φυσικό αέριο στο μέλλον θα είναι και το καύσιμο που θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των ανανεωσίμενων. Γι' αυτό το φυσικό αερίο ε, θα πληγεί από τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ευελιξία έτσι ώστε ο τομέας του φυσικού αερίου να μπορέσει να αντιδράσει και να, προσαρμοστεί στη διείσδυση αυτή των ανανεώσιμων. Εδώ στο, στο μέσον Connecting Europe ε, δεν νομίζω ότι θα ε, καλυφθούν όλες οι απαιτήσει. Θα πρέπει όμως να δοθεί μια όθηση για επενδύσεις ή για έρευνα εκεί όπου δεν υπάρχει εμπορική βιωσιμότητα ή εμπορική αξία έτσι ώστε να μπορέσουν να εσωτερικεύσουν αυτούς τους αριθμούς οι αγορές αλλά ως προς το δίκτυα διαβίβασης για τα επόμενα 8 χρόνια έχουμε 100 δις που προαπαιτούνται, άρα οτιδήποτε ανακύψει από το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη θα είναι πιο αναλογικό. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τα ιδιωτικά κεφάλαια έτσι ώστε να καλύψουμε τα, τις τιμολογήσεις. Θα πρέπει όμως αυτές οι επενδύσεις να γίνουν αποδοτικές. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει και το TNT καθώς και η ανάλυση κόστους ωφελίας. Για να δούμε σχέδια κοινού ενδιαφέροντος στο νέο πακέτο υποδομών. Ε, ελπίζω να μην παρέλειψα κάποιον ή κάτι αλλά όπως είπε και η πρόεδρος, η γνωμοδότηση είναι διαθέσιμη, δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα ακόμα γιατί θα θέλαμε να τη σκεφτείτε και οτιδήποτε θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε και διμερώς. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ τον ε, ε, τον κύριο Ποτότσνικ και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Όλα τα στοιχεία έχουν αποσταλεί. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην ε, έκθεση Χολ. Στην έκθεση της κυρίας Hall, η οποία έχει και το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τα γιοταχή είναι υπεύθυνα για 12% των εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κανονισμός αυτός αφορά το πώς θα επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε ήδη συμφωνήσει για το 2020. Το χρονοδιάγραμμα έχει μεγάλη σημασία, όχι μόνο γιατί πρέπει να περιορίσουμε τα αέρια θερμοκηπίου, κάτι πηγόντος, αλλά έχει και οικονομική σημασία γιατί είναι πολύ καλύτερο για τον κλάδο, τη βιομηχανία, να έχει μια σταθερή πορεία από το να τους ζητάμε να κάνουν ξαφνικά μεγάλες περικοπές. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε, οπότε πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μειωθεί το διοξίδιο του άνθρακα με τρόπο ευέλικτο και που θα στηρίζει την ε, βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία. Είμαι διατεθειμένη λοιπόν να προτείνω δύο αρχές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι έγκαιρες και σοβαρές υπερικοπές και πρέπει να προσφέρουμε στη βιομηχανία μια βεβαιότητα και ευελιξία στο μέλλον. Υπήρξαν 123 τροπολογίες που ε, έχουν εστιαστεί σε 5-6 θέματα. Για αυτά λοιπόν θα μιλήσω. Πρώτα απ' όλα στόχους του 2025. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες από τα 60 γραμμάρια ως τα 75 γραμμάρια για το 2025 και πρέπει νομίζω να βρεθεί μια μέση λύση. Είναι σαφές πως ε, θα μειώνονται οι εκπομπές, θα υπάρξει ένα στόχο του 2025 και είναι σημαντικό η βιομηχανία να έχει κάποια ένδειξη και κάποια βεβαιότητα όσον αφορά το σχεδιασμό. Οπότε ε, και οι κάτι προγραμματίζουν για το 2025, οπότε ε, ούτως ή άλλως το σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, αλλά πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, να γίνουν κάποιες αναθεωρήσεις για να λάβουμε υπόψη τις τεχνολογικές και οικονομικές εξέλιξεις. Κάποιοι λένε να περιμένουμε το νέο κύκλο δοκιμών. Δεν συμφωνώ. Η αυτοκινητομηχανία είναι ε, μέρος της διαδικασίας αναθεώρησης του κύκλου δοκιμών και ξέρει το τι θα γίνει. Και αν περιμένουμε θα έχουμε μεγαλύτερη αβεβαιότητα, καθώς αναμένοντας την νέα Κομισιόν ξέρουμε πως θα έχουμε καθυστερήσεις. Οπότε το να περιμένουμε τον νέο κύκλο δοκιμών σημαίνει πως δεν δίνουμε κανένα νέο μήνυμα. Για τον κύκλο αυτό λοιπόν Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Κάποιοι λένε πως πρέπει να περιμένουμε στο 2021 και υπάρχουν αυτοί που λένε να γίνει νωρίτερα το 2016. Θεωρώ πως καλό θα είναι να ε, συμφωνήσουμε με την Κομισιόν. Λένε πως θα το έχουν έτοιμο το 2014 και χρειάζονται μετά κάποια χρόνια για να γίνει η εφαρμογή. και η μετάβαση από τον υφιστάμενο κανονισμό. Εάν λένε λοιπόν 2017, ας τους πιστέψουμε. Και ας μείνουμε στο 2017. Περνώντας τώρα στις ε, υπερπιστώσεις. Ε, κάποιες επεκτείνονται. Ε, υπάρχουν τροπολογίες που λένε να το διαγράψουμε, άλλες να το επεκτείνουμε. Εγώ θέλω κάποια ευελιξία. Το σαφές είναι πως για να γίνουν οι μεγάλες αλλαγές που πρέπει να κάνουμε τις μεγάλες περικοπές δηλαδή σε εκπομπές, χρειάζονται σταδιακέ αλλαγέ. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο στο τι γίνεται παραδείγματο χάρη με ένα λεγνητικό σταθμό. Υπάρχει ένα όριο και στο τι γίνεται με τον κινητήρα εσωτερική καύση. Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε σε μια νέα τεχνολογία και άρα η επιμηχανία χρειάζεται στήριξη. Το ζήτημα λοιπόν είναι πω εάν έχουμε απεριόριστες τέτοιε πιστώσει θα εξασθενήσει ο στόχος. Και θα έχουμε παραδείγματο χάρη ε, το ζήτημα με τις προτάσεις των Γερμανών συναδέλφων του ΕΛΚ είναι πως ο στόχος ε, θα αυξηθεί κατά 14 ε, γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και ο στόχος παραδείγματος χάρη του 2020 θα πάει στα 109. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι να αλλάξουμε το στόχο, τον αριθμητικό στόχο, αλλά να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το νούμερο. Το αντίστοιχο και με το σκεπτικό αποθήκευση των πιστώσεων αυτών, δηλαδή να τις δώσουμε τώρα που δεν τις χρειάζεται η βιομηχανία και να μπορεί να τους, ε, να τις αποθηκεύσει για να τις χρησιμοποιήσει το 2020. Μα δεν θα βοηθήσει. Αυτό και δεν είναι κίνητρο. Κάποιες τροπολογίες όπως είπα είναι τελείως διαφορετικές, μιλάνε για μια ευέλικτη εντολή και εδώ πέρα το σκεπτικό είναι, ορίζεται ένα όρια, εγώ είπα δύο γραμμάρια, οι σοσιαλιστές είπαν τέσσερα και λέμε πως εάν κάνουν κάτι παραπάνω οι κατασκευαστές, τότε μπορούν να έχουν ένα πιο γενναιόδωρο στόχο. Εάν όμως δεν κάνουν τώρα αυτή την αλλαγή και δεν θέλουν να περάσουν σε ε, ε, νέες ε, τεχνολογίες πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα με τους υφιστάμενους κινητήρες. Και βεβαίως αυτό είναι ένα κίνητρο, αλλά βεβαίως δεν υποβαθμίζει τελείως τον στόχο. Παρακάτω τώρα. Κάποιες άλλες ε, τροπολογίες αφορούν την παρέκκληση χαμηλού όγκου. Υπάρχει μια τροπολογία των κυρίων Φόρντ και Τρεμπεζίνα για να αυξηθεί ο στόχος. Μα δεν έχω πρόβλημα γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο δεν υποβαθμίζει κατά πολύ τον στόχο. Έχει μικρό αποτέλεσμα αλλά δεν μας ανησυχεί. Και βοηθά την βιομηχανία το ίδιο και με τις παρεκκλήσεις ε, των μικρών αγορών. Να αναφερθώ λίγο στην οικοκαινοτομία και την παράμετρο της κοινή ωφελία. Αναφέρθηκε η οικοκαινοτομία, αλλά εγώ αντιλαμβάνω πως είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και πρέπει να γίνει μέσω της επιτροπολογίας. Οπότε θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν την άποψή της. και για την πλευρά της ε, κοινή ωφελία. Τι χρησιμοποιούμε, το βάρος του άνθρακα, το αποτύπωμα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και τα δύο θεωρώ εγώ αμέσως. Επίσης μπορούμε να πάμε στο αποτύπωμα μετά το 2020 καθώς η Κομισιόν ε, προτείνει πως κάτι τέτοιο θα ήταν το λογικό. Είμαι ανοιχτή λοιπόν στις συζητήσεις. Είχαμε ήδη μια καλή συνάντηση νομίζω με τους οδησίγητες και αναμένω τις δικές σας τις απόψεις για να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους για να βρούμε μια ικανοποιητική λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τρία λεπτά έχει τώρα το λόγο ο συνάδελφος Μπρασίνα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, συντάκτρια για την προσπάθεια που έκανε για να επικοινωνήσει με τους κοιόδης εισηγητές και μάλιστα είμαι σε θέση να συμφωνήσω μαζί της όσον αφορά ε, τους ε, γενικούς στόχους για το 2020. Επίσης ανησυχώ για τον τρόπο με τον οποίο διοργανώνεται η δοκιμή του νέου, μάλλον ο νέος κύκλος δοκιμών καθώς και Είμαι βέβαιος πως ε, η ανάφλεξη θα ακολουθηθεί από άλλο ε, σύστημα ε, και ότι θα είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτό όμως στο οποίο διαφωνούμε είναι το θέμα του super credit. Εγώ θεωρώ πως αυτό είναι ένα κίνητρο για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών η εισηγήτρια Όμως η συγγήτρια βλέπει πως εδώ φαίνεται να υπάρχει ένα παραθυράκι για να αποφευχθούν οι κινητήρες χαμηλής εκπομπής ε, διοξιδίου του άνθρακα. Δεν νομίζω πως είναι ουδέτερος ούτε οι άλλες επιλογές, γιατί βασικά ε, μιλούν για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για πιο ευέλικτες, ε, ευέλικτα στάνταρ και στην ουσία ζημιώνονται οι παραγωγοί οι οποίοι δεν δίνουν αρκετό μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων κάτω από το κατόφλι των 35 ε, γραμμαρίων. Άσχετα με το αν τα αυτοκίνητα αυτά είναι ήδη στην αγορά, αν δίνουν ε, καλή, αν μάλλον έχουν ε, προσφέρουν καλή επιλογή τιμή για το χρήστη. Κάτι ακόμα το οποίο είμαι αντίθετο, είναι το, γενικότερα το θέμα των μακροπρόθεσμων στόχων μετά από το 2020. Γιατί πιστεύω ότι όποια και αν είναι ε, η κατάσταση στην ουσία και, και κινούμαστε γύρω από τους στόχους και δημιουργούμε αστάθεια στην αγορά. Και η εισηγήτρια συμφωνεί πως η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αρκετά καλή θέση ώστε να μπορέσει να αντέξει μια ε, ριζική προοπτική στόχων μετά το 2020 για να μπορέσει να τους απορροφήσει. Αυτή τη στιγμή πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες, ε, μάλλον αυτοκινητοβιομηχανίες σε κερδοφόρες βρίσκονται μόνο εκτός της Ευρώπης. Ας σκεφτούμε λοιπόν τις θέσεις απασχόλησης και το ε, δυναμικό των Ευρωπαίων αυτοκινητοβιομηχανών όταν εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το έγγραφο. Αυτή νομίζω ότι είναι η κύριη τομής όπου κατατέθηκαν τροπολογίες και προσβλέπω στην ε, μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Φαν ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για μια καλή έκθεση και για τις προσπάθειες που έκανε να έρθει σε επαφή με τους κοιόδης εισηγητές και νομίζω πως είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε και τις επόμενες εβδομάδες. Στόχος όλων είναι να καταλήξουμε σε κάτι καλό. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή, αυτού του είδους η νομοθεσία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μεγάλες ε, ιδεολογικές ε, αντιπαλότητες. Δηλαδή ο ένας υπερασπίζεται τη βιομηχανία, ο άλλος το περιβάλλον και οδηγούμαστε σε σύγκρουση. Μα δεν χρειάζεται να συγκρουστούμε καθόλου. Αφετηρία είναι το κλίμα και σημαίνει πως πρέπει οι άνθρωποι να εκπέμουν λιγότερα. Οπότε ε, αυτό συνδυάζεται νομίζω με τη στήριξη της ε, βιομηχανίας, της βιομηχανίας του μέλλοντος. Νομίζω λοιπόν πως ε, μπορούμε να βρούμε κάποια κοινά σημεία διακομματικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφωνία πλέον για το ότι οι στόχοι του 2020 είναι θετικοί, εφικτοί και πρέπει να επιτευχθούν και άρα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσαρμοστεί και αυτή η νομοθεσία για να μην εξασθενήσει και έρχομαι άρα στο δεύτερο και σημαντικό το οποίο συζητάμε, κάποια πράγματα δηλαδή που μας απασχόλησαν. Δηλαδή το ότι πρέπει να ορίσουμε νέους, το αν πρέπει να ορίσουμε νέους στόχους για το 2025 ή όχι. Εγώ θα έλεγα πως πρέπει να το κάνουμε, αλλά, αλλά με την απαραίτητη ευελιξία Δηλαδή, εάν ε, πάει πιο γρήγορα η τεχνολογία ή αν υπάρξει κάποιο backloading, ε, αν προκύψει και νέος, και νέος ε, κύκλος δοκιμών, για να υπάρχει και μία ασφάλεια προγραμματισμού για τη βιομηχανία. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για τις περίφημες super credits, τις πιστώσεις αυτές. Πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε πρώτα απ' όλα μεταξύ μας ποιος είναι ο στόχος μας. Όλοι πρέπει να παραδεχτούμε πως τα υφιστάμενες super credits δεν είναι αποτελεσματικές και χρησιμοποιούνται για να ε, υπονομευτεί ε, το πνεύμα της νομοθεσίας. Δηλαδή είναι ένα καλό σύστημα, αλλά δεν είναι σε θέση ε, και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε ε, τη δημιουργία παραθύρων ε, και του ανταγωνισμού. Και τελειώνω κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ πως υπάρχουν διάφορες προτάσεις και εγώ έκανα μια πρόταση, τώρα δεν είναι τίποτα η Αγία Γραφή. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια σε τεχνολογικό επίπεδο να δει με την Κομισιόν ποιο είναι το καλύτερο σύστημα και να προσπαθήσει έτσι να ε, βρει ε, ε, ένα, καλό συμβιβασμό. Οπότε, τι θέλω να πω. Τα super credits πρέπει να υπάρχουν για να προωθηθεί η καινοτομία, όχι για να δημιουργηθούν νέα παραθυράκια για να εξασθενίζουν οι στόχοι που έχουμε. Ευχαριστώ το Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δεν θα ήθελα να επαναλάβω πράγματα που έχουν προαναφερθεί από τους συναδέλφους. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, διότι κατέβαλε πραγματικά μεγάλες προσπάθειες να φτάσουμε σε ένα κοινό παρονομαστή ...παρά την ε, πληθώρα απόψεων που έχουν εκφραστεί και ιδιαίτερα όσον αφορά τις αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, ορισμένες ιδέες είναι εξαιρετικές επί χάρτου, αλλά όχι και στην ε, πράξη. Όταν μιλάμε για επιτάχυνση του εξυγχρονισμού, θα πρέπει να ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα πολλές φορές ε, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο και οι δαπάνες μπορεί να είναι τεράστιες. Συμφωνώ ότι οι στόχοι του 2020 έχουν ε, εισαχθεί σε τέτοιο επίπεδο που είναι δύσκολο για τις αυτοκινητοβιομηχανίες να μπορέσουν να ανταποκριθούν δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσουμε όμως στόχο για το 2025. Μιλάμε για 12 ε, χρόνια αργότερα και συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας μέχρι τότε, γιατί 12 χρόνια είναι πολλά και είναι δύσκολο να ε, θέτουμε φιλόδοξους στόχους για τόσα χρόνια μετά. Συμφωνώ λοιπόν με τους ε, συναδέλφους που θεωρούν ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για 2016-2017. Ας δούμε πώς θα έχουν οι τεχνολογίες εχμής ε, μέχρι τότε ως προς τις ε, υπερπιστώσεις, θεωρώ ότι μπορούν να είναι ευεργετικές για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που θα μπορέσουν να προωθήσουν νέες ιδέες. Γι' αυτό ας ε, δεχτούμε τα super credits ως έχουν, ας μην δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ανασφάλεια στην αγορά. Νομίζω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ μας για πολλές θέσεις εργασίας, γι' αυτό ας μην θέσουμε σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή μας αυτοκινητοβιομηχανία. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τους σκιώδεις. Τώρα ο κύριος Κράμερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τη Φιώνα Χολ για τη γνωμοδότηση αυτή. Να αναφερθώ τώρα σε κάποιες ε, τροπολογίες. Κοιτάξτε, δεν ε, αμφισβητείται ο στόχος του 2020, ειδικά δε όσον αφορά την ε, ασφάλεια της αυτοκινητομηχανίας, πρέπει να αναγνωρίσουμε τους κύκλους των προϊόντων. Δηλαδή τα οχήματα τα οποία θα βγουν στην αγορά το 2020 σχεδιάζονται σήμερα. Δεν, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Πρέπει λοιπόν πάντα να λαμβάνουμε υπόψη πως έχουμε τις πιο φιλόδοξες διατάξεις για το διοξίδιο άνθρακα του πλανήτη. Έτσι. Αν δείτε το τι γίνεται στην Ιαπωνία, στη Νότια Κορέα και στη ΣΥΠΑ, έχουμε αυτή τη στιγμή ό,τι πιο φιλόδοξο υπάρχει. Και βεβαίω δεν είναι όλες μας οι επιθυμίες υπέρ της βιομηχανίας. Καμιά φορά την απειλούμε κιόλα. Και θέλω να πω κάτι το οποίο ε, έχω πει κάποιες φορές. Οι χαμηλότερες εκπομπές στο μέσο όρο του στόλου δεν σημαίνουν αυτομάτως εμπορική επιτυχία. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό οι πρωταθλητές του διοξιδίου του άνθρακα είναι αυτοί που έχουν τι μεγαλύτερε δυσκολίε. Αυτοί οι οποίοι φτάνουν πολυτελή και μεγαλύτερα μοντέλα και πολύ αποτελεσματικά, είναι πιο ανταγωνιστικοί, αλλά ταυτόχρονα έχουν δυσκολίε να επιτύχουν του στόχου. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να δούμε το όριο μεταξύ κίνητρου, κινήτρου και καψονιού, τιμωρίας. Οπότε δεν είναι δυνατόν σήμερα σε τουρκικό παζάρι, που είναι αυτή η συναλλαγή μεταξύ μας, να γράψουμε το τι θα γίνει μετά το 2020. Έτσι. Δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε καμία ιδέα το τι θα γίνει, τι κινητήρες θα υπάρχουν, αν θα είναι ηλεκτρικοί. Δεν είναι τώρα η στιγμή ε, να βγάλουμε ένα νούμερο έτσι, αυθαίρετα επειδή είμαστε πολιτικοί και να πούμε 60-70 γραμμάρια οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να γίνει αργότερα τη στιγμή που πρέπει. Ευχαριστώ Λάγκεν, ευχαριστώ. Το 2008 ήμουν εισηγητής και τότε είχα περάσει τον μακροπρόθεσμο στόχο απέναντι στην ε, αντίσταση γαλλικής και γερμανικής κυβέρνησης και ο στόχος αυτός ήταν κίνητρο για την αυτοκινητοβιομηχανία για να κινητοποιηθεί και να μειώσει το διοξίδιο του άνθρακα. Και θέλω να διαφωνήσω με την κυρία Χολ όταν λέει πως στην ΕΠΑ υπάρχει ο στόχος της μείωσης κατά 5%. Η Καλιφόρνια που είναι η πιο φιλόδοξη έχει το 2011 μέσο στόχο 11,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Εμείς έχουμε στόχο το μισό από αυτό έτσι, μην λέμε ψέματα και δυσκολεύουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία, κυρία Χολ εδώ πέρα. Ε, μαθαίνω δε ότι στην ε, συνάντηση των σκιωδών μαθαίνω πως δεν καλέσατε την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία αλλά την Toyota. Ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, για να έρθω τώρα στην ουσία μόλις τώρα ε, συμφωνήσαμε και παραφέρεται ως πρόταση αυτό το οποίο δεν πέρασε πουθενά ούτε από το Κοινοβούλιο, ούτε από το Συμβούλιο, ούτε στον ε, τριμερή διάλογο. Τώρα, ο κύκλο των δοκιμών. Χρειάζεται ένα ενιαίος κύκλο δοκιμών διεθνώ. Πρέπει να γνωριστούν ε, επίση οι τεχνολογίε. Πρέπει να έχουμε σταθερότητα για τη βιομηχανία όσον αφορά δε τα super credits, την οικοκαινοτομία και την προσπάθεια να δούμε το αποτύπωμα αντί για την μάζα. Αυτή είναι πραγματικά μια επιτυχής πρόταση την οποία είχαμε κάνει ε, τότε και τώρα προσπαθείτε ξανά να μας κάνετε ε, ε, μια προπαγάνδα της Greenpeace. Θεωρώ πως το σχέδιο αυτό έκθεση δεν θα επιτύχει. Η πρόταση της Κομισιόν είναι καλύτερη γιατί στοχεύει σε μια μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ατενίζοντας το μέλλον, σε σχέση με τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα ε, για τα νέα επιβατικά η στοχοθέτηση είναι ζωτική σημασίας. Όμως, η ε, στόχοι μας για το 2020 τονίζει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να κατασκευάσει αυτοκίνητα που να ε, παράγουν ε, χαμηλότερο διοξίδιο του να εκπέμπουν χαμηλότερο διοξίδιο του άνθρακα. Θα πρέπει όμως ε, να κρατήσουμε στάση αναμονής και να δούμε πώς θα εξελιχθεί ένας κύκλος δοκιμών για την παγκόσμια τάση που διαγράφεται ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, γιατί χωρίς αυτές τις ε, πληροφορίες ίσως λάβουμε λάθος αποφάσεις και ίσως είναι καλύτερα να κρατήσουμε στάση αναμονής για να είμαστε σίγουροι. Γιατί μπορεί να επέλθει σύγχυση διαφορετικά και αστάθεια. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να ε, αλλάξει τη στάση, μάλλον να άρει την εμπιστοσύνη της αυτοκινητοβιομηχανίας, με συγχωρείτε. Ε, όσον αφορά την έκθεση αυτή, θα πρέπει να διερευνήσουμε τις δυνατότητες αντικατάστασης ε, της τρέχουσας προσέγγισης, όπου συσχετίζουμε μόνο τις εκπομπές ε, με την κατασκευή ε, με μία προσέγγιση κύκλου ζωής. Έτσι θα λαμβάναμε υπόψη τις εκπομπές ε, αερίων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των αυτοκινήτων, κάτι το οποίο θα έδινε μία πληρέστερη εικόνα της εξελικτικής ε, πορείας των αυτοκινήτων. Ως προς τα πιστοτικά υπερμόρια, μιλάμε για 50 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο και αυτό μέχρι το τέλος του 2015. Και βλέπουμε ότι από τα 3,5% φτάνουμε στο 1,5%. Από το 23% αναφέρεται ότι ό, όταν ε, τα αυτοκίνητα είναι κάτω από τα 35 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, τότε θα λαμβάνουν τα επιστοτικά υπερμόρια. Όμως υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του 16 και το 19 και, πλήρως, και πρότεινα την πλήρωση αυτού του χάσματος. Και τέλος, θα πρέπει να άρουμε τον ε, ύψιστο αριθμό αυτοκινήτων ε, που μπορούν να λάβουν πιστοτικά υπερμόρια γιατί αποτελούν μοχλό μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα, κάτι το οποίο είναι ευεργετικό για το περιβάλλον και, αυτή, ε, και αυτό το σωρευτικό ανώτατο όριο θα ήταν ένας περιορισμός. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι και οι δύο προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης. Μειώνοντας τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, γνωρίζουμε καταρχήν ότι αυτός ο στόχος είναι η τη σημασίας όταν μιλάμε για μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων. Ε, θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής. Αυτό το κριτήριο της ε, χρησιμότητας αυτή τη στιγμή ε, μιλάμε για όγκο. Έχουμε την παράμετρο του όγκου ως προς τη χρησιμότητα. Αν δούμε όμως ε, τον αριθμό των επιβατών, των κινητήρα, τη χρήση του οχήματος και την κατανάλωση ανά χιλιόμετρο, όλα αυτά τα κριτηρία σωρευτικά είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να δούμε και τις ε, διαστάσεις του αυτοκινήτου σε όλα αυτά. Ποιο είναι το μήκος, ύψος, πλάτος και ούτω καθεξής, ε, γιατί έχει μεγάλη σημασία και που αποθηκεύεται αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη η Κομισιόν ως εναλλακτική παράμετρο. Οι μικροί κατασκευαστές ε, που παράγουν μικρά επιβατικά οχήματα ε, ίσως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πολλές φορές ε, έχουμε μεγάλα οχήματα με μεγάλη υποδύναμη και δεν χρειάζονται αυτή την αδειοδότηση την πιστοποίηση, διότι μπορούν να καταβάλουν το αντίτιμο του οχήματος έτσι κι αλλιώς. Και όσον αφορά τη μόλυνση και τη μείωση της μόλυνσης, αυτό είναι και το πιο δυσχερές. Ε, μιλάμε για μικρομόρια, για ηχορύπανση και όχι μόνο για εκπομπές διοξίδιου του άνθρακα. Και όταν κανείς προσπαθεί να καταπολεμήσει μία ε, μορφή ε, μόλυνσης, ας πούμε, ως προς την ηχορύπανση, μπορεί αυτό να έχει άλλα, ε, άλλο εμπλεκόμενο κόστος, άλλο ενεχόμενο κόστος. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά την, κατά κατασκευή και τον κύκλο ζωής. Ως προς τα πιστοτικά υπερμόρια θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα διότι επιτρέπουν τον ανταγωνισμό και θα ρίνουμε και την έρευνα για πλέον καινοτόμες τεχνολογίας Τέλος, ως προς τον υπολογισμό του διοξιδίου του άνθρακα σε συνάρτηση με τη μάζα, ως προς τα γραμμάρια ή το αποτύπωμα γενικότερα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ορισμένους στόχους για την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι το 2020 τα οχήματα θα ζυγίσουν 80 κιλά ε, λιγότερο από ότι τα ε, οχήματα που κατασκευάζονται σήμερα. Και εδώ μιλώ για τα ελαφρά οχήματα. Και βεβαίως πολλές φορές μπορούμε να έχουμε διαφορετική χρήση μετάλλων, τα οποία μπορεί να είναι πιο παχιά ή πιο λεπτά μέταλλα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να ε, παράγουμε ε, λιγότερη, να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια και διοξίδιο του άνθρακα και γι' αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις της Επιτροπής του 2014 που θα είχαν επιπτώσεις και μέχρι το 20. Τι η αξιολόγηση αντικτύπου θα λάβει υπόψη και τις ε, τεχνολογικές αλλαγές που θα επέλθουν. Και δεύτερον, ως προς τα πιστοτικά υπερμόρια, φαίνεται ότι υπόκεινται σε ένα πολυσχηδές ε, ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα υπερμόρια αυτά θα πρέπει να ε, τονίζουν την καινοτομία και το νέο, την κατασκευή νέου στόλου αυτοκινήτων. Πολλές φορές ε, οι καταναλωτές δεν μπορούν να αγοράσουν νέα οχήματα, ενώ τα παλαιά μολύνουν περισσότερο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, μεταχειριστούμε, θα διαχειριστούμε και το θέμα της ταξινόμησης. Μερτσάρος. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μαζί με τους συναδέλφους του ΕΛΚΑ έχουμε υποβάλει πολλές τροπολογίες στην εκθεσία αυτή με στόχο να γίνει κάπως πιο καλή η πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε αυτές. Με την υιοθέτηση αυτού του κανονισμού πρέπει να προστατεύσουμε και την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας μας, γιατί παραμένει εξαιρετικά δύσκολο το περιβάλλον ε, στην Ευρώπη τον Ιανουάριο η ζήτηση νέων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 8,7% φτάνοντας σε ένα ιστορικό χαμηλό ε, από το 1990. Οι ετήσιες αγορές έχουν μειωθεί τα τελευταία 5 χρόνια και έχουμε φτάσει στα χειρότερα επίπεδα των τελευταίων 20 ετών. Οι στόχοι που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ φιλόδοξοι και πολύ περισσότερο στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό τα αυτοκίνητα να παραμείνουν πρόσιτα, οπότε δεν θα πρέπει να το βλέπουμε μεμονωμένα το θέμα αυτό. Οπότε υποστηρίζω το να μην αλλάξουμε την, ε, τους προτινόμενους στόχους για το 2020. Από την άλλη ο κανονισμός αυτός αφορά τους στόχους του 2020. Κατά την άποψή μου λοιπόν δεν πρέπει να θέσουμε ενδεικτικούς στόχους για μετά το 2020 αυτή τη στιγμή συμφώνω με τις ε, τροπολογίες δε που έχουμε καταθέσει, θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα αυτό το 2017 το νωρίτερο. Η βιομηχανία λοιπόν χρειάζεται μια βεβαιότητα και πρέπει να συνεχίσουμε βεβαίως να μειώνουμε την κατανάλωση καυσίμων ε, προς το συμφέρον και των καταναλωτών μας. Αλλά το να θέσουμε ένα στόχο για μετά το 2020 χωρίς να γίνει πρώτα η σωστή διαδικασία δημιουργεί περισσότερη αβεβαιότητα καθώς τα νούμερα αυτά θα είναι αυστηρά πολιτικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, κανόνες προβλέψιμους και με ε, αποτελέσματα βιώσιμα. Ρέμπεκ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι σκιώδης στην έκθεση αυτή, ούτε μιλάω εξ ονόματος ολόκληρης της ομάδας μου, της Γκουε, γιατί ε, δεν ξέρω αν θα είμαστε ενωμένοι εδώ πέρα αλλά ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ομάδας μου θα ζητούσε κάποια μετριοπάθεια θα έλεγα γιατί τα αυτοκίνητα ως ένα φαινόμενο που σχετίζεται με τον εκδημοκρατισμό της ε, κοινωνίας βελτιώνει την κινητικότητα των ανθρώπων αλλά ακόμα και τις δυνατότητες αναψυχής για ευρύτατα τμήματα της κοινωνίας. Από την άλλη, το αυτοκίνητο έχει και άλλες πτυχές. Και η αυτοκινητομηχανία βεβαίως προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας, γιατί υπάρχουν και πολλοί υπεργολάβοι, ε, υποκατασκευαστές. Ε, εκεί πέρα είχαμε πάρα πολλές απώλειες λοιπόν θέσεων εργασίας ε, και δεν ανάγκη να επιδεινώσουμε την κατάσταση αυτοκινητομηχανείς δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή και οι υπεργολάβοι τους, παραδείγματος χάρη στην Τσεχία, όπου ε, η μέση ηλικία των αυτοκινήτων είναι πάνω από 14 έτη. Ε, είναι καλύτερα στη Δυτική Ευρώπη, αλλά στην Ανατολική είναι χειρότερα τα πράγματα. Τι θέλω να πω λοιπόν. Ε, έχει ήδη αναφερθεί. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να αγοράσει καινούργια αυτοκίνητα. Και οι νέες τεχνολογίες τα κάνουν πιο ακριβά συνήθως. Βεβαίως, εάν είναι να απαγορεύσουμε τη χρήση των παλαιότερων αυτοκινήτων ε, και αυτό δεν θα είναι δημοκρατικό. Θα περιορίζουμε έτσι τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας μας. Ποιος μπορεί να αγοράσει αυτοκίνητο κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Να μην μιλήσω για τα εκτός δρόμου που κάνουν 100.000-150.000. Βεβαίως αυτοί που αγοράζουν αυτά τα αυτοκίνητα δεν επηρεάζονται από την κρίση. Αυτά. Συμφωνώ δε με τους κύριους... Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει να παρέμβει. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχολεία σας. Ήδη σχολιάσαμε το σχέδιο έκθεσης και γι' αυτό θα, θα αναφερθώ στα θέματα που αφορούν τις ε, τροπολογίες. Ε, υπάρχουν τροπολογίες όσον αφορά τα υπερμόρια που δίνονται δυνατότητα, όπως είπε και ο εισηγητής, να, πετυχ... να επιτευχθούν οι στόχοι. Δεν είμαστε υπέρ εξαιρετικά γενναιόδωρων τέτοιων ε, ε, σχεδίων. Ιδιαίτερα πρέπει να μπορέσουν να μπουν και οι τράπεζες, ε, γιατί έτσι θα καθυστερηθεί η επίτευξη των στόχων του 2020. Κάποιες άλλες τροπολογίες που προτείνουν ε, τη θέσπιση ορίων για τα υπερμόρια θα πρέπει να αυτά να μπορούν να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις, να δίνουν κίνητρα, χωρίς όμως να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων. Σε σχέση με τον κύκλο δοκιμών, η Κομισιόν έχει ε, ήδη θεσπίσει μια διαδικασία που θα αρχίσει να ισχύει από το 2014 για την καταγραφή και των εκπομπών. Είναι σημαντικό λοιπόν για τους καταναλωτές. Πιστεύουμε πως δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσει η εισήγηση του νέου, της νέας διαδικασίας ε, ε, δοκιμών. Επίσης στις προτάσεις μας έχουμε φροντίσει ότι η προσαρμογή από τον ισχύοντα κύκλο δοκιμών στον επόμενο δεν θα απαιτήσει εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια από τους κατασκευαστέ. και αυτό είναι σαφές και από την πρόταση και θα πρέπει να καθησυχάσει τους ε, κατασκευαστές. Και έπειτα να σας αναφέρω και την ε, αναθεώρηση μετά το 2020 γιατί σε πολλές τροπολογίες ε, συνδέονται με την αναθεώρηση του 2020. Η Κομισιόν ε, θέλει να δώσει βεβαιότητα σχεδιασμού στους κατασκευαστές. 12 χρόνια νωρίτερα λοιπόν έχουμε θεσπίσει αυτή την ημερομηνία. Το 2017 σημαίνει πως η σχετική νομοθεσία θα υιοθετηθεί μόνο το 2019 και δεν θα έχουν χρόνο να προσαρμοστούν οι κατασκευαστές. Γι' αυτό και προτείνουμε η αναθεώρηση να γίνει το 2014. Και τέλος έγινε μια ερώτηση από τον εισηγητή σε σχέση με τις καινοτομίες. Οι διαδικασίες είναι ανοιχτέ σε αναθεώρηση. Εμείς συνεργαζόμαστε με τους ενδιαφερόμενους φορείς και αναζητούμε ικανοποιητικές λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. γιατρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα έλεγα πως ε, ήταν πολύ καλό που άκουσα όλα αυτά τα σχόλια. Υπάρχει μια γνήσια συνένεση ότι δεν θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τους στόχους του 2020. Αυτό ήταν σαφές. Η βιομηχανία ζητά ε, βεβαιότητα ε, και γι' αυτό θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Θα ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα ένα επικοδομητικό σχόλιο του κ. Τοσανόφσκι για αυτή την μεγάλη συζήτηση για τα υπερμόρια, είναι ευέλικτη εντολή, ό,τι και να το πούμε αυτό. Εγώ νομίζω πως θα πρέπει να μείνουμε στην πρόταση της Κομισιόν και θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αν δεν υπάρχει συνένεση για τις τροπολογίες, θα ήταν ε, καλύτερο να δεχτούμε την πρόταση της Κομισιόν από αυτού για τους στόχους του 2025. Όλοι συμφωνούμε πως θα πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα σχεδιασμού. Θα ήθελα ωστόσο να δοθεί ένα σαφές μήνυμα προς τη βιομηχανία ότι υπάρχει μια κατεύθυνση, ότι το χρόνο δεν πρέπει να εκπλαγούν όταν η Κομισιόν θα υποβάλει κάποιους ε, αυστηρότερους στόχους από όσους έχουμε τώρα. Προσεκτικά λοιπόν να διατυπώσουμε ότι ό,τι και αν πούμε τώρα είναι πολιτικές ενδείξεις προς μια κατεύθυνση και μόνο του χρόνου θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα ε, ενώ θα έχουμε, αφού μάλλον θα έχουμε και την ε, μελέτη αντικτύπου και όλα τα στοιχεία από την Κομισιόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδες εισηγητές. Ήδη έχουμε κάνει μια συνάντηση των σκιωδών που ήταν βοηθητική κάνουμε και μια ειδική συνεδρίαση ε, για το ευέλικτο σύστημα όπου καλέσαμε και τους ενδιαφερόμενους φορείς για να δουν πώς λειτουργεί το σύστημα στην Καλιφόρνια και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις και όλους τους συνεργάτες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χόλ. 19 Μαρτίου προβλέπεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή και περνάμε στο τελευταίο σημερινό, μάλλον σημείο της πρωινής σημερινής διάταξης. Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Ο συνάδελφος Πίπερ δεν είναι εδώ. Τον αντικαθιστά ο συνάδελφος Λάγκε, ο οποίος θα έχει και το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Πίπερ μου ζήτησε να παρουσιάσω την πρότασή του. Ευχαρίστω θα το κάνω γιατί πριν από δύο χρόνια ήμουν συγητή στην Επιτροπή Βιομηχανίας για το θέμα αυτό και γνωρίζω τα σχετικά προβλήματα. Έχουμε λοιπόν τον στόχο των 147 γραμματείου που πρέπει να διατηρηθεί, αλλά βεβαίω πρέπει να δούμε και το εφικτό του πράγματος και αυτό το υποστηρίζει ο κύριος Πίπερ και θεωρεί πως πλην μερικών εξαιρέσεων ε, για τι οποίε υπάρχουν τροπολογίε και αφορούν τον κύκλο δοκιμών, ε, της διατάξεις ε, για τυχόν απαλλαγές. Θεωρεί λοιπόν πως μπορεί να υποστηρίξει την πρόταση της Κομισιόν. Συνολικά υπάρχουν 54 ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, η πλειοψηφία από την κυρία Φανμπρέμπτ ε, και τους ε, πράσινους δείχνουν αυτές, όπως δυστυχώς και τα τελευταία χρόνια και στην έκθεση ΦΟΛ, μικρή επαφή με τις ιδέες που έχουμε εντός της Επιτροπής μας. Οπότε, ε, μιλάνε για μια αυστηροποίηση από τις 147 στα 128 μέχρι και 110 γραμμάρια, χωρίς κάποια αιτιολόγηση για το γιατί πρέπει ε, να αλλάξουν οι στόχοι που υιοθετήσαμε πριν από δύο μόλις χρόνια. Ο κύριος Πίπερ, ε, πόσο βλέπω, είναι κατά. Κατόπιν ε, για το 2025 ο στόχος 85 μεταξύ, μεταξύ 85 και 110 γραμμαρίων δεν έχει καμία λογική. Τα δε μικρά αυτά φορτηγά είναι το εργαλείο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αν κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα θα δημιουργήσουμε προβλήματα όχι μόνο για τους κατασκευαστές αλλά για τους χρήστες. Όταν έχουμε δηλαδή τεράστια έξοδα εξοπλισμού. Αυτό κατά την άποψή μου και την άποψη του κυρίου Πίπερ δεν είναι λογικό. Και αυτή η φανταστική αριθμή επίσης είναι πάλι αυθαίρετη. Δεν υπάρχει κάποια βάση, κάποια αξιολόγηση αντικτύπου. Είναι απλά προτάσεις της Greenpeace. Να μειωθούν αυτά τα σούπερ μόρια. Αυτή είναι η πρόταση των σοσιαλδημοκρατών και των πρασίνων είναι ένα σημαντικό κίνητρο για τους κατασκευαστές. Δεν πρέπει να καταργηθούν. Ανταυτού ε, οι σοσιαλδημοκράτες, η, η σκιώδης ε, συγγήτρια των σοσιαλδημοκρατών λέει να υπάρξει κάποιος καταναγκασμός. Δηλαδή, αν δεν ε, επιτυγχάνει κάποιο ε, ποσοστό της αγοράς ε, να τιμωρείται ο κατασκευαστής. Μα είτε έχουμε κίνητρο, είτε έχουμε τιμωρία. Αλλιώ είναι τα πράγματα τελείω λανθασμένα και βλάπτουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και ειδικά, όπω σα είπα, τι μικρομισέ επιχειρήσει. Μετά προτείνεται να μπουν κόφτε ταχύτητα. Έγινε η συζήτηση στην Επιτροπή Μεταφορών. Δεν είναι συζήτηση δική μα και δεν ταιριάζει σε αυτή την έκθεση. Ε, εγώ προσωπικά ε, θέλω να σας πω πως ε, εντάξει μπορούμε να βάλουμε κάποιες επιπλέον περιορισμούς σαν μικρά φορτηγά αλλά δεν ταιριάζει σε αυτήν εδώ πέρα την νομοθεσία και ειδικά σας πω πως ειδικά στο φάκελο αυτό ας είμαστε μετριοπαθείς μην το παρακάνουμε και θέλω να παρακαλέσω εξ ονόματος του κυρίου Πίπερ να ακολουθήσουμε μια λογική γραμμή Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις. Καταρχήν η κυρία Βαν Μπρέντε. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη, γιατί έδωσα πολλά, πολλά επιχειρήματα στην νομοθεσία ΚΑΖ. Ε, είναι παράλληλα τα πράγματα, έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για τα super credits και για τον κύκλο δοκιμών και για το ε, στόχο 20-20-20 και σε αυτή την επιτροπή λοιπόν πρέπει να δούμε τους δύο φακέλους ε, παράλληλα. Η συζήτηση είναι παράλληλη με αυτό το οποίο έγινε για τα αγιοταχή. Ίσως είναι η στιγμή να ξαναγίνει μια συζήτηση. Δηλαδή να λέμε πως όλες οι τροπολογίες είναι κακές ε, δεν είναι τακτική αυτή. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Για να πετύχουμε κάποιους στόχους για τα super credits. Ε, εντάξει, δεν είναι και η Αγία Γραφή, έτσι. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Ε, υπάρχουν και άλλες προτάσεις άλλων πολιτικών ομάδων. μπορεί να απτυχθεί νομίζω ένα σύστημα νομίζω για τα ελαφρά φορτηγά και τα αυτοκίνητα. Με στόχο τον ίδιο δηλαδή καινοτομία α, αλλά τι να σας πω και τους στόχους του 2020 εμείς τους θέσαμε. Δεν είναι τόσο ε, άσχημη η κατάσταση, απλά προσπαθούμε να έχουμε φιλόδοξους στόχους και χωρίς να έχουμε παραθυράκια μετά για τη βιομηχανία. Να συζητήσουμε αν θέλετε τεχνικά. Θεωρώ πως η τεχνογνωσία της ε, Κομισιόν ε, για το Super Credits μπορεί εδώ πέρα να μας ε, χρησιμεύσει. Εγώ δεν είμαι ειδική στο θέμα. Αλλά πρέπει να γίνει συζήτηση δεύτερον. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά τώρα σε σχέση με τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά, γιατί η στόχη για τα αυτοκίνητα είναι πιο φιλόδοξη νομοθεσία. Οπότε πρέπει να σημειωθεί και εδώ πέρα κάποια πρόοδο. Τελειώνω κυρία Πρόεδρε. Για τον κόφτη στα λεωφορεία. Εντάξει δεν κολλάει εδώ πέρα. Αλλά υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα στον περιορισμό των εκπομπών δεξιού του άνθρακα. Και πρέπει να το δούμε και εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Κράμερ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν ε, νομίζω από εμά τροπολογίες στην ε, έκθεση Πίπερ. Ε, δεχόμαστε αυτά τα οποία έχει προτείνει και δικαίω σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα με τα ελαφρά φορτηγά υπάρχει μια πιο έντονη συζήτηση για το στόχο του 2020 αλλά θέλω να υπενθυμίσω πως αυτό το νούμερο, το 147 ε, γραμμάρια, το ορίσαμε πριν από δύο χρόνια με δύσκολη συζήτηση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό. Οπότε μόνο αυτό μας λέει ότι δεν πρέπει να το ξανανοίξουμε τώρα. Χρειάζεται και μια ασφάλεια προγραμματισμού α, ε, για τη βιομηχανία, γιατί τα φορτηγά έχουν ακόμη μεγαλύτερο κύκλο σχεδιασμού και παραγωγής από τα γεωταχή. Εγώ Προσωπικά συμφωνώ με τον κύριο Πίπερ πως τα super credits εδώ πέρα έχουν νόημα όπως και στα γεωταχή αλλά είμαι πεπισμένος πως έχει πιο νόημα να έχουμε περισσότερα super credits εδώ πέρα από τις γεωταχή γιατί υπάρχει ε, εδώ πέρα μια αγορά πιθανή για ηλεκτρικούς κινητήρες, ε, ε, για τις εταιρείες που έχουν στόλους και κάνουν αστικές μεταφορές και θα μπορούν π.χ. να δημιουργήσουν ε, είτε ε, καταστάσεις με μπαταρίες είτε καταστάσεις φόρτισης. Και το επιχείρημα τώρα να ορίσουμε στόχους για το 2025 είναι αυτό που ανέπτυξα πριν για τα αυτοκίνητα. Και μην ξεχνάτε πως έχουμε πολύ μικρότερη βάση δεδομένων από ό,τι στα Ιωταχή και υπάρχουν ε, το θέμα των διαφόρων πλατφορμών, πάρα πολλά πράγματα δεν ξέρουμε λοιπόν το τι θα γίνει ε, και το πώς θα μετρηθούν και δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν έχουμε στοιχεία για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Δεν είναι λοιπόν η στιγμή αυτή τη στιγμή να ε, λέμε νούμερα ε, εκ νέου. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να ορίσουμε μακροπρόθεσμους στόχους. Ο κύκλος δοκιμών ισχύει ότι και για τα ταχύ. Δεν είναι ικανοποιητικός ο υφιστάμενος κύκλος γιατί δεν είναι πρακτικός. Αλλά ε, σημασία έχει η τυποποίηση του κύκλου αυτού. Και αυτό ισχύει και για τα γεωταχή. Πρέπει να υπάρξει ένας κύκλος ε, ο οποίος ε, θα είναι πρακτικός και αυτός πριν κρίνουμε τα νέα νούμερα, γιατί θα αποτελέσει βάση του υπολογισμού. Δεν μπορεί τα νούμερα να τα ορίζουμε πολιτικά, αλλά μαθηματικά. Και το ζήτημα είναι να έχουμε περισσότερο χρόνο. Οπότε πρέπει πρώτα να καταλήξουμε στον κύκλο δοκιμών. Οπότε υποστηρίζουμε αυτό το οποίο έχει κάνει ο κύριος Πίπερ και παρακαλώ να το κάνετε κι εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο ε, Κράμερ, ο κύριο Κοζανόφσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. και εγώ, όπως και ο σκιώδης των Ευρωπαίων Συντηρητικών και ε, μεταρρυθμιστών θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση Πίπερ και νομίζω ότι τα ε, πιστοτικά υπερμόρια τάσσονται υπέρ της καινοτομίας ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, γιατί αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν καινοτομίε που υπηρετούν αυτό το σκοπό. Γι' αυτό νομίζω ότι τα όρια εκπομπών τα συμφωνήσαμε μετά από μακρά συζήτηση και δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να αλλάξουν. Ε, συναντήθηκα με τον κύριο Πίπερ, ε, συμφωνώ με την εργασία του, τον υποστηρίζω και πιστεύω ότι θα πρέπει να τιμήσουμε την εργασία του, γιατί εδώ μιλάμε για βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα αυτό μπορούμε να το κάνουμε έμπρακτα με αυτόν τον τρόπο. Vidal Κουάδρας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κανονισμός αυτός ε, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Καλωσορίζουμε την επιβεβαίωση της Επιτροπής για τους στόχους του 2020 147 τα γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Είναι εφικτός ο στόχος και θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, αυτοκινητοβιομηχανία έτσι ώστε να, να γίνουν ε, οι κατάλληλες αλλαγές. Συμφωνώ με τον κύριο Πίπερ ότι αυτή η στόχη ε, για το 2020 που προκαθορίστηκαν το 2011 είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη πριν ορίσουμε στόχους για μετά το 2020, θα πρέπει να κρατήσουμε στάση αναμονής, όπως είπα και προηγουμένως. Να δούμε πώς θα ε, ολοκληρωθεί ο κύκλος δοκιμών για την εναρμόνιση του του κύκλου για την εναρμόνιση της αντιμετώπισης των ε, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, εξετάσει αυτή την προσέγγιση και να δούμε, την, να προωθήσουμε την προσέγγιση του κύκλου ζωής των οχημάτων. Η Επιτροπή θέλει κάτι να μας πει. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τα σχόλια, με όσα ελέγχθησαν για τα πιστοτικά υπερμόρια και τον κύκλο ζωής καθώς και τους στόχους μετά το 2020, θα ήθελα να πω τα εξής. Ε, έγινε λόγος για ε, περιορισμό ταχυτήτων, περιοριστές ταχυτήτων και θεωρώ ότι είναι ένα από τα μέσα που θα ήθελε να εξετάσει η Επιτροπή και να διερευνήσει για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να το ε, παρεκτείνουμε και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε σχέση με τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο. Ε, Λάγκε. Ναι, εξ του κυρίου Πίπερ θέλω να πω πως ενδιαφέρεται πάρα πολύ στο να καταλήξουμε σε μια ως το δυνατόν ευρύτερη συμφωνία. Υποθέτω πως θα κάνει τις ανάλογες συζητήσεις. Αλλά όσον αφορά τους στόχους ε, και μετά τη συζήτηση δεν νομίζω να προέκυψε λόγος να ορίσουμε στόχους για το 2025. Υπάρχει ο στόχος των 147 γραμμαρίων όπως πρότεινε η Κομισιόν και έτσι πρέπει να παραμείνει. Και τα 147 γραμμάρια είναι ο στόχος των ΙΠΑ το 2025 για τα απλά ΙΧ που είναι ο δικός μας στόχος του 2020 για τα μικρά φορτηγά. Έτσι. Για τα ΙΧ 5 χρόνια αργότερα. Οπότε μην τρελαθούμε εδώ πέρα. Είναι φιλόδοξος ο στόχος και τα μικρά φορτηγά ε, δεν είναι μόνο θέμα βιομηχανικής πολιτικής αλλά και μικρομισών επιχειρήσεων. Αυτές θα χρησιμοποιούν. Ευχαριστώ, συνάδελφε Λάγκερ. Προβλέπετε ψηφοφορία στις 19 Μαρτίου στην Ήτρη και εμείς έχουμε ραντεβού εδώ στις 3. Καλή σας όρεξη.